Αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα. Όλοι έχουμε λάβει την ημερήσια διάταξη για τη σημερινή συνεδρίαση. Αν ε, δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, μπορούμε να την υιοθετήσουμε ως έχει. Διερμηνία παρέχεται σε 18 γλώσσες σήμερα. Η συνεδρίαση μεταδίδεται στο διαδίκτυο συνήθως. Και όλα τα έγγραφα σας έχουν διατεθεί σε ηλεκτρονική μορφή. Σημαντικό είναι ότι πρέπει να εγκρίνουμε τα πρακτικά μια σειρά συνεδριάσεων προηγουμένων, συγκεκριμένα της 24ης και της 28ης Νοεμβρίου, της 1ης Δεκεμβρίου και της 5ης Δεκεμβρίου του 2016. Εάν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, μπορώ να θεωρήσω ότι εγκρίθηκαν τα πρακτικά. Uh, uh, Μπορούμε να προχωρήσουμε στη συζήτηση. Όπως γνωρίζετε, έχει ολοκληρωθεί το σχέδιο έκθεσης ε, τον ε, Δεκέμβριο. Αποτελείται από τρία μέρη. Ε, το μέρος που περιγράφει τα γεγονότα όπου δεν μπορούν να υποβληθούν τροπολογίες, το σχέδιο συστάσεων όπου μπορούν να υποβληθούν τροπολογίες και, και επίσης ε, το σχέδιο συμπερασμάτων. Και μπορούν ε, <clears throat> να υποβληθούν τροπολογίες ε, κατά το υπόλοιπο της εντολής της Επιτροπής μας. Μία ώρα και 50 λεπτά προβλέπονται για τη συζήτηση αυτή και θα δώσω πρώτα το λόγο στους εισηγητές, τον κύριο Κίζα και πρώτα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την εισαγωγή αυτή. Εύχομαι σε εσά και στους ε, όλα τα καλά για το 2017. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις πολιτικές ομάδες για την εξαιρετική συνεργασία. Καταφέραμε να ε, εκπονήσουμε ένα πολύ ισορροπημένο τμήμα της έκθεσης που αναφέρεται στα γεγονότα. στο περιγραφικό κομμάτι καταφέραμε να καταλήξουμε σε συμβιβασμό που μπορούν να δεχτούν ε, όλες οι πλευρές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Κέρμπεν Γιάν Κερμπράντη καθώς και όλους τους άλλους ε, σκιώδεις εισηγητές. Και η γραμματεία, θα πρέπει να τονίσουμε, έκανε εξαιρετική δουλειά και μας βοήθησε πολύ κατά τη διάρκεια των ε, διαπραγματεύσεων. Θα ήθελα πολύ να συνεχίσουμε αυτήν την επικοδομητική συνεργασία. Το αντικειμενικό κομμάτι της ε, έκθεσης επιτρέπει στον καθένα να υποβάλει συστάσεις. Από πλευράς ε, του ΕΛ και βλέπω να υπάρχουν τα εξής κεντρικά σημεία. Ε, κατά τις ακροάσεις δεν διαπιστώσαμε κανένα φταίξιμο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχουν ε, πολύ μεγάλες διαφορές ανάμεσα στην ε, μέτρηση των οξυδίων ε, του αζότου στα εργαστήρια κατά τις δοκιμές και στις πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Αυτό είναι γνωστό εδώ και αρκετό καιρό και είναι δύσκολο να καταλάβουμε γιατί απαιτεί τόσο χρόνο να εφαρμοστεί η νέα μέθοδος δοκιμών. Είδαμε ότι ε, το φταίξιμο δεν είναι αποκλειστικά της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής, ε, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πίεσε για την προώθηση του νέου κύκλου δοκιμών. Κατά τη διάρκεια των ακροάσεων διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης σε επίπεδο κρατών μελών. Πρέπει να βελτιωθεί η δουλειά εντός των κρατών μελών. Και θα πρέπει να είναι σαφές σε ποιο κράτος μέλος ε, είναι αρμόδιο για την έγκριση τύπου. Ε, αν ε, από ένα άλλο κράτος μέλος όμως υπάρξουν υποψίες, είναι δεμένα τα χέρια του λόγω των κανόνων της ενιαίας αγοράς. Υπάρχει εδώ λοιπόν περιθώριο βελτίωσης. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει καλύτερα να εποπτεύουν την έγκριση τύπου και να έχουν καλύτερη εποπτεία της αγοράς. Ε, σχετικές ε, προτάσεις βελτίωσης ε, έχουν υποβληθεί. Και θέλουμε να υποστηρίξουμε τις προσπάθειες αυτές με τις εργασίες μας. Τέλος, θα ήθελα να μιλήσω για το μέλλον της τεχνολογίας diesel. Η τεχνολογία αυτή στην Ευρώπη είναι πολύ διαδεδομένη. Στο πλαίσιο της ε, ευρωπαϊκής πολιτικής ε, για την καταπολέμηση της ε, αλλαγής του κλίματος έχει κεντρικό ρόλο. Θέλουμε να πετύχουμε χαμηλότερες τιμές εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και με την χρήση των σωστών τεχνολογιών θα μπορέσουμε να τηρήσουμε και τα χαμηλά επίπεδα εκπομπών οξυδίου του αζότου. Πιστεύουμε ότι αυτά αποτελούν καλά νέα για την Ευρώπη. Σας ευχαριστώ και πάλι για την καλή συνεργασία και ελπίζω να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την ε, επικοδομητική συνεργασία. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στο δεύτερο εισηγητή, τον κύριο Γκεπράντη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω ευχαριστώντας τον συνεισηγητή μου, τον κύριο Γιάννης ε, Γκίζικε, και τον προκάτοχό του, τον Παύλο Ζόλμπα. Ε, όλοι γνωρίζουμε ότι όταν ε, ψηφίσαμε για την σύσταση της Επιτροπής αυτής, ακολουθήσαμε διαφορετικές προσεγγίσεις και πλευρές, αλλά τελικά ήταν άκρος καρποφόρες συζητήσεις. Πάρα πολύ καλή συνεργασία. Είμαι άκρος ικανοποιημένος με το σχέδιο εκθέσεως που έχετε μπροστά σας αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι κατορθώσαμε να συντάξουμε ένα πολύ καλό κείμενο, πιστικό περιεχομένο, πιστική έκθεση. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους ιδιαίτερος τους και όσοι ηγητές, κυρίως για τα στοιχεία που παρουσιάσαμε έπρεπε να ε, συμφωνήσουμε επ' αυτών γιατί δεν τροποποιείται το κείμενο ούτε σε επιτροπή ήταν πολύ συνεργατική η στάση όλων των σκιωδών και έτσι ε, ήταν άκρος καρποφόρο το αποτέλεσμα όσον αφορά την παρουσίαση των στοιχείων. Σημαντικότατη αυτή η βάση. Αυτό δείχνει ότι ε, λειτουργήσαμε ως ε, Εξεταστική Επιτροπή με συνεκτικό τρόπο και θα πρέπει να δούμε πώς θα προχωρήσουμε όσον αφορά το τροποποιήσιμο τμήμα του κειμένου. Ο Γένς ήδη ανέφερε κάποια στοιχεία βασιστήκαμε επί του τεράστιου όγκου εγγράφων που λάβαμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και από άλλες πηγές και προφανώς και επί των ακροάσεων. Αυτή ήταν η βάση της εκθέσεως που συζητούμε. Τα συμπεράσματα είναι αρκετά σκληρά. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ακόμα και σκληρά είναι τα συμπεράσματα για τα κράτη-μέλη. Και αν υπάρχει ένα γενικό συμπέρασμα που μπορεί να συναγάγει κανείς, είναι ότι το σύστημα που δημιουργήσαμε για την έγκριση αυτοκινήτων στην Ευρώπη δεν λειτουργήσε με τον τρόπο που θα θέλαμε. Οι ευθύνες σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο δεν ετηρήθησαν Οπότε είναι σημαντικότατο να τροποποιήσουμε το σύστημα, όπως κάνουμε κυρίως στην Επιτροπή ΙΜΚΟ. Εξετάζοντας το περιεχόμενο της εκθέσεως, θα το διαβάσατε όλοι, διότι δημοσιεύθηκε την εβδομάδα πριν από τα Χριστούγεννα. Δεν φοβηθήκαμε να κατονομάσουμε ε, αυτούς που έχουν ευθύνε. Κατονομάσαμε τα κράτη-μέλη που έπαιξαν ιδιαίτερα αρνητικό ρόλο και κυρίως στην Τεχνική Επιτροπή για τα οχήματα, κυρίως κολλησιεργώντας όσον αφορά τη θέσπιση νέων δοκιμών, επικρίναμε σκληρά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την ευθύνη που έχει, διότι επέτρεψε στα κράτη-μέλη να χρονοτριβήσουν όσον αφορά την εφαρμογή του νέου συστήματος. Η εφαρμογή των μέτρων ήταν κάκιστη στα κράτη-μέλη. Όλα αυτά αναφέρονται στην έκθεση. Κάποιοι από εσά σε ατομική βάση ή σε ομαδική βάση θέλετε να αλλάξετε κάποια τμήματα. Εγώ θα μπορούσα να δεχτώ την έκθεση αυτή και χωρίς καμία τροποποίηση. Αλλά νομίζω ότι σε κάποια σημεία θα μπορούσε να βελτιωθεί. Κυρίως εφόσον έχουμε ακόμα ακροάσεις Έχουμε ακρόαση του Υπουργού Εξωτερικών του, της Σλοβακίας και του Υπουργού μάλλον και τους Ιταλούς θα ακούσουμε και εξακολουθούμε να λαμβάνουμε έγγραφα και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από άλλες πηγές. Πρέπει να προχωρήσουμε στην Επιτροπή και να συναγάγουμε συμπεράσματα, να τα συζητήσουμε και να προχωρήσουμε στις στάσεις. Ευχαριστώ εκ νέου όλους για την άριστη συνεργασία και προσβλέπω στα σχόλια των διαφόρων ομάδων που είναι παρούσες σήμερα. Εγώ ίδιος πρέπει να ζητήσω συγγνώμη, πρέπει να πάω στην Επιτροπή Περιβάλλοντος διότι έχουμε ψηφοφορία στις 9.40 θα αποχωρήσω και θα επιστρέψω, αλλά το προσωπικό μου εδώ θα ακούσει τα διάφορα σχόλια που θα εκφραστούν. Ευχαριστώ. Κύριε Μπράντι, να δώσω το λόγο στους κοιόδης εισηγητές Η κυρία Λονέ, ζήτησε το λόγο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Το είπαν οι δύο συνεισηγητές και τους οποίους θέλω να ευχαριστήσω. Έγινε μια σημαντική συλλογική προσπάθεια πριν από την έκθεση αυτή ε, σε μια πολύ σημαντική φάση της διαδικασίας και βεβαίως απέφερε καρπούς η προσπάθεια αυτή. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν τους συζητητές, τους ε, ε, σκιώδεις αλλά και τη γραμματεία αυτής της Ερευνητικής Επιτροπής ε, που εργάστηκαν σκληρά, όλους τους συμβούλους, τους βοηθούς ε, που μας βοήθησαν. Η ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών ε, είναι ικανοποιημένη από αυτό το σκέλος του κειμένου και θεωρούμε ότι όσο ευρύτερη στήριξη στήχει αυτή η έκθεση στην Ερευνητική Επιτροπή τόσο πιο ισχυρή θα είμαστε στην Ολομέλεια. Πρέπει δηλαδή αυτή η έκθεση να είναι όσο γίνεται πιο ισχυρή και σε ό,τι αφορά τις διαπιστώσεις και σε ό,τι αφορά τις συστάσεις. Πρέπει να μπορέσουμε να επηρεάσουμε το μέλλον των ζητημάτων αυτών που είναι και περιβαλλοντικά και βιομηχανικά αλλά και ζητήματα απασχόλησης. Θελήσαμε λοιπόν να εργαστούμε συλλογικά και όσο γίνεται επικοδομητικά, όπως, είπε ο κ. Γκερμπράντι, θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν τους κύριους συζητητές από, από την FDD, από τους πράσινους, από την ΚΟΕ. Ε, τα αρχικά κείμενα ήταν ήδη καλά, διότι είχε γίνει μια δουλειά με τις ακροάσεις, ε, μια δουλειά ουσιαστική ε, και έτσι υπάρχει μεγαλύτερη σύγκληση στις προτάσεις και στις διαπιστώσεις, αλλά πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Κάποιες ε, προδευτικές προτάσεις δεν μπήκαν στο σκέλος αυτό, αλλά θα υποβληθούν μορφή τροπολογιών στα συμπεράσματα και στις συστάσεις. Θα ήθελα να αναφερθώ σε μια σειρά σημεία που για μας είναι σημαντικά και θα θέλαμε να μπουν ε, στο μέρος με τις διαπιστώσεις. Ε, θα πρέπει να μπορούμε να συμπεριλάβουμε το θέμα της υπέρβασης του διοξείδου του άνθρακα. Δεν υπήρχε βεβαίως ε, στο εμείς, αλλά είναι σημαντικό. Μια αναφορά ε, στην ε, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η έλλειψη εντολής η GRC, του JRC μάλλον από την Κομισιόν, η έγκαιρη γνωστοποίηση του προβλήματος, οι πιέσεις που υπήρξαν από τον κλάδο στα κράτη-μέλη, που στη συνέχεια μεταφέρθηκαν και στο CTVM, η ακρίβεια των παραγόντων συμμόρφωσης και των ΠΕΜΣ που ήταν προβληματική, ε, τα διάφορα συστήματα ακύρωσης, το γεγονός ε, ότι είναι η απαγόρευση σαφής παρότι υπάρχουν κρίζες ζώνες ή ε, λήψη στην εποπτεία της ευρωπαϊκής αγοράς. Θέλω λοιπόν να επαναλάβω αυτό που κ ήρθε η στιγμή τώρα που έχουμε αυτούς τους γάντζους να γαντζώσουμε εκεί τις αρχές μας και να τις αναπτύξουμε. Εμείς θα υποβάλουμε τροπολογίες πριν 18 Ιανουαρίου και για τις συστάσεις και για τα συμπεράσματα. Είναι σημαντικά τα συμπεράσματα διότι ουσιαστικά ανοίγουν την, την τελική έκθεση, όμως οι συστάσεις είναι αυτές που θα μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τα πράγματα. Αν οι συστάσεις δεν είναι στο ύψος των περιστάσεων, τότε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα έχει παίξει το ρόλο του. Και εδώ είναι που μας περιμένουν οι συμπολίτες μας. Περιμένουν συγκεκριμένες προτάσεις. Οι τροπολογίες θα υποβληθούν για να επιμείνουμε σε αυτές τις αδικαιολόγητες προθεσμίες ό,τι αφορά την ανάγκη εποπτείας. Να επενθυμίσουμε τις αδυναμίες της υπάρχουσας νομοθεσίας, την ανεπάρκεια των ακυρώσεων, τις ευθύνης των κρατών μελών αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να επανέλθουμε στην υπερεκπροσώπηση του βιομηχανικού κλάδου στις βιομάδες εργασίας. Όσο πιο ισχυρό είναι το κείμενο στην ομάδα έρευνας, τόσο καλύτερο αποτέλεσμα θα έχουμε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να είναι όσο πιο ενωμένο στο θέμα αυτό, έτσι ώστε οι συστάσει μα να ληφθούν σοβαρά υπόψη. Θα είναι η ευκαιρία να βελτιώσουμε και τι εργασίε των ερευνητικών επιτροπών γενικότερα. Δεν ήταν καλό το χρονοδιάγραμμα, δεν ήταν ιδανικό. Είχαμε και την έκθεση ε, για ε, τα οχήματα και την ε, τυποποίησή τους. Ε, συνεχίζουμε τώρα εντωμεταξύ να τις ακροάσεις ενώ έχει ήδη ε, ολοκληρωθεί η έκθεση Γι' αυτό δεν είναι και τόσο λογικό. Πρέπει επίση σε επίπεδο διαβίβαση εγγράφων να βελτιώσουμε τα πράγματα, σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η μέθοδο εργασία μα πρέπει να βελτιωθεί, διότι είναι προφανέ ότι στο μέλλον θα έχουμε και άλλε τέτοιου είδου ερευνητικέ επιτροπέ. Σα ευχαριστώ όλου για την προσπάθειά σα. Έχουμε ακόμα πολλή δουλειά μπροστά μα. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω επίσης το λόγο σε άλλους συναδέρφους με τη διαδικασία Καρσιά. Ο κ. Πανκολόπης, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Η έκθεση αυτή κατά την άποψή μου κάνει μια ισορροπημένη ε, ανάλυση σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό των εκπομπών στον τομέα της αυτοκινημιομηχανίας έγινε μια κατανομή ευθυνών μεταξύ κρατών μελών και κομισιών με λογικό τρόπο, αλλά το να κατανείμουμε θεσμικά τις ευθύνες δεν ενδιαφέρει τόσο τους συμπολίτε μας. Βλέπουμε εδώ ότι υπάρχει ανάγκη μιας νομοθεσίας πιο ε, ευθυγραμμισμένης και μια πιο αυστηρή εφαρμογή της. Να έχουμε ένα αποτελεσματικό σύστημα κυρώσεων. Χώρες όπως η δική μου, η Ισπανία, ε, καθυστέρησαν ε, τις δοκιμές ε, σε ιδανικές ε, συνθήκες. Ε, αυτό δεν πρέπει να ξαναγίνει, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες επανεργοποίησης. Πάντως, ε, φτάσαμε σε ένα υψηλό επίπεδο συμφωνίας. ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτό. Η πρόσωπός μας και η ε, η ομάδα των, από των Δημοκρατών ε, κάνουν ό,τι, έκανε ό,τι μπορούσε έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα και να μην τα ξαναβρούμε μπροστά μας στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ντάνς. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ όλους εδώ. Προφανώς πλησιάζουμε στο τέλος της διαδικασίας αυτής θα υπάρξουν ευκαιρίες και αργότερα, αλλά νομίζω και σήμερα είναι πολύ καλή ευκαιρία να ευχαριστήσουμε τους συνεισηγητές και τους κοιόδες εισηγητές για όλη τη δουλειά που έχουν κάνει πάνω στο θέμα αυτό. Έχουν εμπλεκεί πολύ στην εργασία αυτή. Έχει γίνει πολύ σκληρή δουλειά για την εκπόνηση της ε, έκθεσης αυτής ε, και έπρεπε να εξεταστούν όλες οι σχετικές πληροφορίες. Η Κριστίν μίλησε για το χρονοδιάγραμμα. Και αυτή είναι μία από τις συστάσεις μας. Έχουμε τώρα ακροάσεις ε, μετά από την ολοκλήρωση της έκθεσης. Ε, δεν ξέρουμε ε, αν θα πέσει καμιά βόμβα, κάτι πολύ σημαντικό δηλαδή που δεν θα συμπεριληφθεί στην έκθεση. Αλλά μαθαίνουμε και νομίζω ότι οι εμπειρίες μας εδώ θα είναι πολύ χρήσιμες κατά την εκπόνηση κανόνων για μελλοντικές εξεταστικές επιτροπές. Η έκθεση αυτή αναφέρεται στο τι πήγε στραβά ε, και εντοπίζει αυτούς που δεν έκαναν αυτό που έπρεπε όσον αφορά τους ε, κανόνες ε, για τις εκπομπές ε, οχημάτων. Καταρχάς, οι εθνικές αρχές δεν εφήρμοσαν σωστά τους κανόνες και τις σχετικές κυρώσεις. Επίσης, δεν υπήρχε αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς, κάτι που αντίκειται στο ενωσιακό δίκαιο. Και παρά τη μεγάλη διαφορά των εκπομπών στο εργαστήριο και ε, τον δρόμο. Ε, ήταν γνωστό από το 2010 και παρόλα αυτά κανένα κράτος μέλος δεν ασχολήθηκε, ε, δεν εξέτασε δηλαδή ε, αν συμμορφώνονται τα οχήματα που κυκλοφορούν στους δρόμους του με τους κανόνες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούσε και θα έπρεπε να είχε κάνει πολύ περισσότερα για να αντιμετωπίσει την κατάσταση όσον αφορά τις συνθήκες οδήγησης γιατί καθυστέρησε τις δοκιμές RDE τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι η τεχνολογία υπήρχε εδώ και πολλά χρόνια. Γιατί δεν έδωσε συνέχεια ε, στην ε, επικοινωνία ανάμεσα στην ε, JRC και τη, τα, τις δικές της υπηρεσίες. Και το Κοινό Συμβούλιο Ερευνών. Ε, μάθαμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προχώρησε περαιτέρω διότι θεώρησε ότι μπορεί να υπάρξουν ε, ότι μπορεί να υπάρχει χρήση των ε, συστημάτων αναστολής από τους παρασκευαστές, το οποίο είναι πολύ λάθος το ότι δεν έκανε κάτι. Και ενώ οι κατασκευαστές ε, αναφέρονται στα βαρέα οχήματα όσον αφορά τις εκπομπές, ε, δεν αναφέρονται στα ελαφρά οχήματα και αυτό θέτει πολλά ερωτηματικά. θα πρέπει να φροντίσουμε να μην ξανασυμβεί αυτό για να έχουμε νέες εξεταστικές επιτροπές ε, σε 20-30 χρόνια. από Στη δική μου χώρα δεν ε, ε, είναι πολύ ωραίο να λέει κανεί ε, αυτή τη στιγμή ότι η απάντηση είναι περισσότερη Ευρώπη, αλλά νομίζω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση χρειάζεται. Χρειαζόμαστε ανεξάρτητες δοκιμές ώστε να μην κάνουν τα στραβαμάτια οι εθνικές αρχές και αυτό θα είναι καλό όχι μόνο για τη δημόσια υγεία αλλά και για τον ανταγωνισμό. Για να διασφαλίσουμε αυτή την ανεξαρτησία η ευρωπαϊκή εποπτεία θα πρέπει να πραγματοποιείται μέσω νέου οργανισμού που θα είναι αρμόδιος για την εποπτεία της αγοράς. Αν θέλουμε να μάθουμε από τις καλύτερες πρακτικές, ας κοιτάξουμε στις Ηνωμένε Πολιτείε και, την, και τον ε, Οργανισμό Προστασίας του Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Πολιτειών, ε, χωρίς τον οποίο δεν θα βρισκόμασταν εδώ σήμερα η ευθύνη για την ποιότητα του αέρα και οι εκπομπές των οχημάτων ε, δεν θα πρέπει να είναι θέματα χωρισμένα ανάμεσα σε δύο γενικές διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που συχνά έχουν ε, αντίθετους στόχους. Θα πρέπει λοιπόν από την DG Grow να ε, μεταφερθεί το σχετικό χαρτοφυλάκιο στην Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή η έκθεση αυτή. Νομίζω ότι όλες οι πολιτικές ομάδες μπορούν να είναι ε, περήφανες για αυτήν και ελπίζω οι συνάδελφοι από την Επιτροπή ΙΜΚΟ να υιοθετήσουν τις συστάσεις μας ε, όταν ψηφίσουν για το θέμα της έγκρισης τύπου αργότερα εντός του μήνα αυτού. Πιστεύω ότι ω Κοινοβούλιο μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τη δουλειά που έχουμε κάνει στην Επιτροπή αυτή και να είμαστε περήφανοι για τη δουλειά όλων των συναδέρφων πάνω στο θέμα αυτό. Χαίρομαι που μπορώ να σας πω ότι η έκθεσή μας αποτελεί πολύ καλή βάση για την περαιτέρω συζήτηση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Ντάνς. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Έιβη, τη σκιώδη εισηγήτρια. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θέλω να συμφωνήσω με αυτά που λένε οι συνάδελφοι. Κατά την άποψή μου αυτή η έκθεση είναι πολύ καλή. Ευχαριστώ τους συνεισηγητές που έκαναν αυτή τη δουλειά. Τα συμπεράσματα μα συμφωνούν, ευρέω συμφωνεί. Έπρεπε να εντοπιστούν οι ευθύνε σε περιπτώσει κακή ε, αντιμετώπιση του θέματο από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κρατών μελών. Θα ήθελα να πω όμω ότι είναι κάπως αμφίσιμο το κείμενο όσον αφορά τις ευθύνες των παρανόμων αυτών μηχανισμών αναστολής όπως αναφέρεται στο σημείο 4. Κυρίως όσον αφορά την παράκομψη των αδύναμων ίδιων ε, κανόνων περί των δοκιμών. Όσον αφορά τον έλεγχο και την ε, έγκριση των αυτοκινήτων έχουν ευθύνες οι αρμόδιες αρχές. Από την άλλη πλευρά, μόνο σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει υποψία για την παρανομία των στατικικών που ακολούθησαν οι κατασκευαστές των αυτοκινήτων ή συμμορφωθούν την νομοθεσία. Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα ήταν χρήσιμο ε, να αναφέρουμε την ύπαρξη πριν τη θέσπιση του Euro 5 και του Euro 6 και άλλων δοκιμών εργαστηρίων πολύ καλύτερων που θα μείωναν δραστικά τις εκπομπές που επιτρέπονται κατά τη διάρκεια της έγκρισης τύπου αυτών των αυτοκινήτων θεωρώ το κομμάτι που καθορίζει τις μελλοντικέ ευθύνες αδύναμο όσον αφορά τη χορήγηση έγκρισης και τη διάθεση στην αγορά και τον έλεγχο της αγοράς. Θα έπρεπε να τονίσουμε περισσότερο τη δυνατότητα να αναθέσουμε τους ελέγχους συμμόρφωσης στην υπηρεσία σε τρίτο φορέα, όπως ψηφίσαμε και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Όσον αφορά το παράγοντα συμμόρφωσης, θα πρέπει να ζητήσουμε ρητά την μείωση, διότι όλες οι μαρτυρίες που ακούσαμε και κάποιες ε, αποδείξεις και δοκιμές με τα ΠΕΜΣ έδειξαν τη δυνατότητα να σεβαστούμε ήδη τους, ε, τα όρια στους δρόμους. Όσον αφορά τις δοκιμές συμμόρφωσης σε λειτουργία, σε υπηρεσία, θα ήταν καλό να δώσουμε διακριτική ευχέρεια στις αρχές όσον αφορά ποιες δοκιμές θα γίνονται και πώς θα διεξάγονται και όχι να τις περιορίζουμε την ελευθερία. Τέλος προσθέτω ότι πιστεύω ότι χρειάζεται να συμπεριλάβουμε την δημόσια πρόσβαση στα αποτελέσματα των ερευνών που διεξάγονται από τα κράτη-μέλη και να επενθυμίσω ότι θα μπορούσε να είναι χρήσιμο να επαναλάβουμε την ανάγκη να εγγυόμεθε την παρουσία και των μικρών ομάδων στις, επιτροπές, στις εξεταστικές επιτροπές. Ευχαριστώ για τη δουλειά που έγινε και σίγουρα αυτό είναι ένα σημαντικό έγγραφο που ελπίζω να μπορέσει να υπερψηφίσει το Κοινοβούλιο με μεγάλη πλειοψηφία. Ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο στον κύριο Ερντούκ. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους. Ε, θα ήθελα να ε, συμφωνήσω με αυτά που είπε ο, ο συνάδελφος ο κύριος Ντάνς. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους ε, δύο συνεισηγητές καθώς και τους σκιώδεις συνεισηγητές. Ε, θετικά με εξέπληξε το πως η έκθεση αυτή έχει συνοψίσει όλες τις επικρίσεις που έχουν ακουστεί ε, στην Επιτροπή μας. Ε, αρχικά είχα την εντύπωση ότι μετά τις συζητήσεις που ακούσαμε το τελευταίο δεκάμινο αυτό δεν θα είναι πολύ εύκολο, αλλά εκτιμώ το πόσο έχει γίνει αυτό με αντικειμενικό τρόπο. βρίσκω πολύ θετικό το πόσα θέματα έχουν συμπεριληφθεί ε, στην έκθεση. Η Εξεταστική Επιτροπή έχει ε, κάνει σημαντική δουλειά και έχει διαπιστώσει τι λήψεις υπήρχαν κατά την μέτρηση των εκπομπών και κατά την έγκριση τύπου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη στο παρελθόν θα μπορούσαν ε, ενωμένοι να ε, αποτρέψουν κάποιες ε, πρακτικές. Χαίρομαι πολύ που όλα αυτά λοιπόν παρουσιάζονται στην έκθεση. Θα ήθελα να επαναλάβω ότι η, έκθεση, ότι η Επιτροπή μας δεν στρέφεται κατά συγκεκριμένων κατασκευαστών ή συγκεκριμένων χωρών κράτη-μέλη όμως ε, και η βιομηχανία θα πρέπει να βγάλουν ε, τα σωστά συμπεράσματα ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Η Επιτροπή μας ε, λοιπόν έχει πετύχει πολλά, έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Ευχαριστώ όλους όσους συμμετείχαν στις εργασίες και προσβλέπω σε καλή συνέχιση των εργασιών στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και για να πάμε στον κύριο Βάντερ Κάμπ για να ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε λέει ο Νομίζω ότι φτάσαμε στο τέλος του ευχολογίου για το νέο έτος. Τέλος πάντων, ευχηθώ ξανά ευτυχισμένο τον καινούριο χρόνο. Έχω ένα κρυολόγημα, αλλά τέλος πάντων ελπίζω να ακουστώ καλά ξεκάθαρα στην παρέμβασή μου. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τους δύο συνεισηγητές και τους σκιώδης συγητές για τη δουλειά που έκαναν. Συνέβαλα, ήμουν παρόν στις περισσότερες ακροάσεις και τις συναντήσεις και οι περισσότερες λεπτομέρειες και συζητήσεις ε, είναι γνωστές σε και τα έγγραφα και όλα αυτά τα είδα. Εξέτασα όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες οι οποίες είναι σημαντικότατες. Διαφωνήσαμε σε κάποια τεχνικά ζητήματα. Καμιά φορά ακουγόταν και κάποια παραμύθια γιατί αναμίχθηκε η αλήθεια με την αναλήθεια, με αναλήθειες σε αυτά που υπόθηκαν. Αυτό που είναι σημαντικό από τη συζήτηση αυτή είναι ότι είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι πάρα πολύ μεγάλη σημασία της. Μέχρι τώρα δεν είχαμε επιπτώσεις, δεν είδαμε κάποιον ε, από τη διοίκηση αυτοκινητοβιομηχανίας να φύγει, ούτε κάποιος επίτροπος να παραιτηθεί. Δεν βλέπουμε να αναλαμβάνεται η ευθύνη από κάποιον. Εγώ θα έλεγα ότι έχω κάπως σοκαριστεί από τον τρόπο με τον οποίο στην Ευρώπη και κυρίως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έγινε η αντιμετώπιση του προβλήματος. Όταν ε, λαμβάνεις μεγάλο όγκο εγγράφων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πολλά ηλεκτρονικά μηνύματα, τότε καταλαβαίνεις ότι κάτι τρέχει, κάτι πάει στραβά και βλέποντα τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων γενικών διευθύνσεων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των διαφόρων εμπλεκομένων φορέων, ε, εγώ βλέπω ότι δεν κάναμε πολύ καλά τη δουλειά μας τα τελευταία δύο χρόνια. Λέω εμείς, διότι πιστεύω ότι και το Ευρωκοινοβούλιο είναι ένα κομμάτι της ε, όλη εικόνα. και μπορούμε να μάθουμε για το μέλλον από αυτό που συνέβη από τη διαδικασία. Ο ρόλο των κρατών μελών. Πολλά υπόθηκαν. Ο κύριος Γκεμπράντι ανέφερε τα βασικά στοιχεία και υποστηρίζω αυτά που είπε. Τι θα κάνουμε τώρα, αυτό είναι το θέμα, Πρόεδρε. Όπως είπε και ο συνάδελφο από το ECR, τώρα τίθεται θέμα δημόσιας υγείας. Αφορά την υγεία των πολιτών μας το ζήτημα. Υπάρχουν τα στατιστικά στοιχεία. Όταν βλέπετε τι συμβαίνει εντός των αστικών ε, χώρων, στο αστικό περιβάλλον, βλέπουμε ότι έχουμε πάρα πολλές ρηπαντικές ουσίες που εκπέμπονται από τα οχήματα και πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση. Εξετάζοντας τη νομική βάση της Επιτροπής μας και τη δομή της Επιτροπής μας, ε, μιλήσαμε κυρίως με προσώπους φορέων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Χρειάζεται να υπάρχει εμπιστοσύνη τελικά στην αυτοκινητοβιομηχανία για να γίνει σωστή δουλειά. Όσον αφορά λοιπόν τη μεγάλη εμπιστοσύνη στην αυτοκινητοβιομηχανία, θέλω να πω ότι με αυτό που συνέβη υπήρξε μεγάλη απογοήτευση. Μετά είδαμε πώς αντιμετωπίστηκε το σκάνδαλο στις Ηνωμένε Πολιτείε και στην Ευρώπη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ε, επευλήθησαν τεράστια πρόστιμα, ε, υπήρξαν συλλήψεις των ε, υπευθύνων των διαφόρων εταιριών που μετά απελευθερώθηκαν. Όμως έγινε κάτι, εν κατακλείδη πρόεδρε. Για μένα δεν είναι πολύ ξεκάθαρο ποιος θα δώσει συνέχεια στις συστάσεις αυτές. Τι θα συμβεί, ποια συνέχεια θα δοθεί θα, θα παραμείνει ένας πυρήνας της Επιτροπής μας με αρμοδιότητα να επαγρυπνεί ούτως ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμμορφωθεί με τις συστάσεις μας. Δηλαδή, ποιος θα φροντίσει να γίνει κάτι, να δοθεί κάποια συνέχεια ε, και να υλοποιηθούν, να ακολουθηθούν οι συστάσεις με επαγγελματικό τρόπο. Εξάλλου, δεν αναφέρομαι μόνο στη νέα νομοθεσία η οποία θα εφαρμοστεί προς το τέλος του 2019, αλλά πιο γενικά, με πιο μεγάλο, πιο μακρινό ορίζοντα, τι θα κάνουμε. Αλλάζουμε θητεία, αλλάζουν οι επίτροποι, όταν αλλάζουν οι θητείες πρέπει να δούμε τι θα γίνει, πώς θα δοθεί κάποια συνέχεια. Θα μπορούσαμε να έχουμε κάποια απάντηση πάνω σε αυτό. Θα ήθελα να καταλάβω ποιο θα μπορούσε να δώσει συνέχεια στην καλή δουλειά που κάναμε μέχρι τώρα σε αυτή την Επιτροπή. Αυτό είναι το θέμα. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο και στους δύο συγητές, ούτω ώστε να απαντήσουν. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ακούσω τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Άννα Σικόφσκα είναι εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επικεφαλής της μονάδας που ασχολείται με τον τομέα των αυτοκινήτων στη Γενική Διεύθυνση Γκρό. Ευχαριστώ Πρόεδρε και καλημέρα σε όλους. Θέλω να ευχηθώ ότι καλύτερο για τη νέα χρονιά σε όλους. Σας ευχαριστώ για το σχέδιο έκθεση και για το σχέδιο συστάσεων καθώς και για το γεγονός ότι δίνετε την ευκαιρία στην Κομισιόν να συμμετάσχει σε αυτή την συνάντηση. Θα ήθελα να κάνω κάποια σύντομα σχόλια. Καταρχήν να υπογραμμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συνεργαστεί με την Επιτροπή αυτή με σε πλήρη διαφάνεια, εκτεταμένα. Σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να το πράττουμε αυτό έως το ολοκληρωθεί το έργο σας. Είναι ο μόνος τρόπος και ο καλύτερος τρόπος για να καλύψουμε όλες τις ανησυχίες, να φτάσουμε στα καλύτερα δυνατά συμπεράσματα και να ε, μπορέσουμε να φέρουμε στο φως όλα τα στοιχεία. Επίσης, αυτή η Επιτροπή κοιτάζει βεβαίως το παρελθόν. Όμως, εξίσου σημαντικό, ίσως και περισσότερο, ε, θα πρέπει να ανοίξει η έκθεση αυτή το δρόμο για το μέλλον. Έτσι λοιπόν αναμένουμε και ελπίζουμε ότι η έκθεση θα αναγνωρίσει την προσπάθεια της Κομισιόν για να δημιουργηθεί το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο όχι μόνο για τις εκπομπές αλλά και για την έγκριση τύπου. Η δουλειά που λαμβάνει η χώρα αυτή τη στιγμή στην ΙΜΚΟ και στην ΕΜΗ συνδέονται. Η Κομισιόν έχει υποβάλει μια πρόταση που έχει τεράστιες δυνατότητες ε, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα κενά και τις αδυναμίες του παρού συστήματος. Ελπίζουμε λοιπόν ότι η έκθεση της ΕΜΙΣ ε, θα ακολουθήσει αυτή την οδό την οποία προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το τρίτο που είναι επίση σημαντικό είναι ότι ελπίζουμε και αναμένουμε ότι η έκθεση αυτή θα βρει το σωστό σημείο ισορροπίας. Όχι μόνο να εντοπίσει τις ευθύνες των μεν και των δε για αυτά που συνέβησαν, αλλά να αναφέρει πού έλαβε χώρα τελικά η απάτη ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τι πρέπει να γίνει στο μέλλον. Και βεβαίως η έκθεση πάει πέρα από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Ε, Υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα θεσμικά που αφορούν και την Κομισιόν. Αυτές οι συστάσεις, αυτά τα συμπεράσματα ε, θα πρέπει να μας οδηγήσουν το να σκεφτούμε σε βάθος τα ζητήματα αυτά και να μπορέσουμε να απαντήσουμε. Είμαστε στη διάθεσή σας ε, για περαιτέρω συνεργασία ε, και για να διαλευκάνουμε οποιοδήποτε απορίες έχετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, είμαστε κοντά στο τέλος της συζήτησης αυτής. Θα πάμε πίσω στους εισηγητές. Ο κύριος Γκίζικε είναι εδώ ακόμα. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τις παρατηρήσεις τους. Ακούσαμε πολλούς επένους, ε, κάτι που με κάνει να αναρωτιέμαι αν όντως τα κάναμε σωστά. Αλλά ιδιαίτερα κατά την εκπόνηση του αντικειμενικού κομματιού, επειδή δεν μπορούσαν ε, να υποβληθούν τροπολογίες, ε, προσπαθήσαμε να πετύχουμε συνένεση ανάμεσα στις πολιτικές ομάδες. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με τον τρόπο αυτό. Όσον αφορά τις επιμέρους ε, παρατηρήσεις των συναδέλφων, ήταν πολύ επικοδομητικέ και υποστηρίζουν τις εργασίες μα. Η συνάδελφο Εύη αναφέρθηκε στα συστήματα αναστολή. Αυτό είναι πράγματι πολύ σωστό διαπιστώσαμε ότι όταν υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες, οι αρμόδιοι λένε ότι θα πρέπει αυτό να το λύσει η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και υπάρχει τότε απλά διαδικασία διαμεσολάβησης και όχι απόφαση. Αυτό είναι πολύπλοκο. Οι κατασκευαστές ε, έχουν εκμεταλλευτεί το περιθώριο που είχαν και γι' αυτό λυπάμαι που δεν θα έχουμε ακρόση με την Όπελ, διότι θα μπορούσαμε να τους ρωτήσουμε σχετικά με το σύστημα που κλείνει ε, σε συγκεκριμένη θερμοκρασία και δεν ε, μετράει πια τις, δεν μειώνει πια τις εκπομπές. Ε, ίσως θα μπορούσαμε να ζητήσουμε από την Όπελ γραπτή απάντηση. Θα θέλαμε περαιτέρω διευκρίνηση δηλαδή πάνω στο θέμα αυτό. Κατά τα άλλα, η συζήτηση ήταν πολύ αντικειμενική και θα ήθελα να παρακαλέσω τον συνάδελφο Ντάνς να μην μπούμε σε πολιτικές λεπτομέρειες. Ε, ήταν πάρα πολύ δύσκολο στην Επιτροπή μας ε, να προσκαλέσουμε τους Επιτρόπους. Ο Επίτροπος Εφερχόγεν ήρθε κατόπιν τεσσάρων προσκλήσεων. Θα πρέπει να αποφύγουμε να με ε, μονομένους ε, επιτρόπους. Εμείς ε, ως Επιτροπή εξετάζουμε την ε, εσφαλμένη ε, συμπεριφορά της Κομισιόν και είμαι αισιόδοξο ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε με αυτό στο μέλλον. βέβαια, συχνά βλέπουμε, ακούμε πολλούς επένους για εκθέσεις εισηγητών και τελικά βλέπουμε εκατοντάδες ανθρωπολογίες. Πιστεύω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε στις βασικές τροπολογίες, να πω ανοιχτά ότι αν έχουμε εκατοντάδες τροπολογίες και προσπαθήσουμε να επανεφεύρουμε τον τροχό, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να διατηρήσουμε αυτή την διάθεση συμβιβασμού. Ο Γκέρβεν Ιαν Γκέρμπραντι είπε πριν ε, και αυτό μου άρεσε πολύ ότι μπορεί να δεχτεί την έκθεση υπό την μορφή που έχει αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν τροπολογίε, αλλά ίσω θα ήταν ε, καλό οι συνάδελφοι να επικεντρωθούν στι βασικέ τροπολογίε, ώστε να πετύχουμε συνενετικό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά τι τροπολογίε. θα σας δώσω το χρονοδιάγραμμα. Ε, η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι 18 Ιανουαρίου 2017 στις 3 η ώρα το απόγευμα. Από Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου, μπορείτε να αρχίσετε να μας τις στέλνετε. Θα τις εξετάσουμε στην Επιτροπή μας ε, στις 9 Φεβρουαρίου και θα ψηφίσουμε στις 28 Φεβρουαρίου και κατόπιν ε, θα έχουμε την ε, συζήτηση στην Ολομέλεια που προβλέπεται για τον Απρίλιο. Προτείνω σύντομο διάλειμμα για να επιτρέψουμε στους ομιλητές για την επόμενη ακρόαση να προσέλθουν. Πέντε λεπτά διάλειμμα. Και θα προχωρήσουμε στην ακρόαση του κυρίου Βίκτορ Στρόμτσεκ, που είναι υφυπουργός του Υπουργείου Μεταφορών στην Σλοβακία. Εντάξει, έτσι.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 Λοιπόν, μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο σημείο τη σημερινή Τετάρτη και θα ακούσουμε τον κύριο Στρότσεκ, που είναι υφυπουργό ε, Περιφερειακή Ανάπτυξη και Μεταφορών τη Σλοβακία. Καλώ ήρθατε, κύριε Στρότσεκ. Ευχαριστούμε που δεχτήκατε την πρόσκλησή μα. Κύριο Στρότσεκ είναι υπουργό από τον Απρίλιο του 2013 και αναμένεται να μας αναφέρει το πώς η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία εκπομπές αυτοκινήτων εφαρμόζεται στη Σοβακία και πληροφορίες για το Εθνικό Σύστημα Εγκρίσεως Τύπου και πώς λειτουργεί σαν εκπρόσωπος της χώρας που ασκεί την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ενώσης ο κ. Στρόμψεκ επίσης αναμένεται να σχολιάσει τη συζήτηση που έλαβε χώρα για το θέμα των εκπομπών, για τη μέτρηση των εκπομπών στο Συμβούλιο των Μεταφορών και τα αναμενόμενα επόμενα βήματα. Με ένα εκατομμύρια οχήματα που παρήχθησαν το 2015, η Σλοβακία είναι η έκτη μεγαλύτερη παραγωγός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεύτερο νέο κράτος μέλος παραγωγός μετά Τσεχική Δημοκρατία και μεγαλύτερος παραγωγός παγκοσμίως κατά κεφαλή. Η Σλοβακία ε, παράγει Volkswagen, PSA, ε, Kia και αναμένεται να ξεκινήσει και παραγωγή Jaguar Land Rover τον επόμενο χρόνο. Ε, η αρχή εγκρίσεως τύπου στη Σλοβακία ανήκει στο Υπουργείο Μεταφορών, Οικοδομών και Περιφερειακής Ανάπτυξης που εκπροσωπεί ο κ. Στρόμτσεκ. Υπάρχουν 10 κοινοποιημένες τεχνικές υπηρεσίες. Η Σλοβακία δεν χορηγεί εγκρίσεις τύπου σύμφωνα με τον κανονισμο 715 κλπ. Να επενθυμίσουμε στα μέλη τα παρόντα ότι έχουν λάβει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τις απαντήσεις στις αρχικές ε, γραπτές ερωτήσεις ε, μπορούν να βρουν το έγγραφο αυτό στο φάκελο της ε, συνεδριάσεως. Έχουμε μία ώρα και 40 λεπτά που προβλέπεται να διαρκέσει η συζήτηση αυτή. Ξεκινάμε λοιπόν με την εισαγωγική δήλωση του Υπουργού και μετά τα μέλη θα υποβάλουν ερωτήσεις σύμφωνα με την αρχή που ακολουθούμε του πινκ-πονγκ. Πολλοί γνωρίζουν. Ο πρώτος γύρος ερωτήσεων υποβάλλει τους συγγητές. Ακολουθεί ένας εκπρόσωπος κάθε πολιτικής ομάδας, ένα πεντάλεπτο ο καθένας. Καλώς. Ο κ. Σόμτσεκ λοιπόν μπορεί να προβεί στα εισαγωγικά του σχόλια και έχει 10 λεπτά στη διάθεσή του. Thank you very much. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ. Καταρχά θα ήθελα να σα ευχαριστήσω θερμά που με προσκαλέσατε στην Επιτροπή σα. Θα ήθελα να ευχηθώ και καλή χρονιά σε όλους. Για μας είναι ιδιαίτερα σημαντική η Επιτροπή σας. Είμαστε, όπως ήδη υπόθηκε, από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές οχημάτων στην Ευρώπη και μάλιστα κατά κεφαλή είμαστε ο μεγαλύτερος κατασκευαστής. Η οικονομία μας εξαρτάται από την βιομηχανία αυτοκινήτων, αντιπροσωπεύει πάνω από το 20% του ΑΕΠ και γι' αυτό χρειαζόμαστε σαφείς κανόνες και θα πρέπει να μπορούμε να εξετάσουμε την ποιότητα των οχημάτων συνολικά. Τα τελευταία χρόνια έχουν ε, αλλάξει τα πράγματα. Στο παρελθόν εξετάζαμε κυρίως ε, το διοξίδιο του άνθρακα, εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα, λόγω της αλλαγής του κλίματος ε, και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισήγαγε οριακές τιμές και οι κατασκευαστές έπρεπε να μειώσουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Το αντίτιμο όμω ήταν η αύξηση των οξυδίων του αζότου. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε μια συνολική λύση για το μέλλον. Όσον αφορά την Προεδρία της Σλοβακίας, ε, η Προεδρία μας ολοκληρώθηκε πριν από δύο εβδομάδες και καταβάλαμε προσπάθειες να βρούμε συστημική προσέγγιση στις ε, διαπραγματεύσεις ε, για τον κανονισμό σχετικά με την έγκριση τύπου που αποτελεί και τον πυρήνα του όλου προβλήματος. Ε, καταφέραμε να πετύχουμε συμφωνία όσον αφορά τα τεχνικά άρθρα κυρίως όσον αφορά την επιστοποίηση συμμόρφωσης και την ε, διευκόλυνση της καταχώρησης ε, παλαιών σειρών. Είμαι πεπισμένος ότι η Σλοβακική Προεδρία πέτυχε ό,τι καλύτερο μπορούσε εντός ε, του χρονικού διαστήματος που είχε στη διάθεσή της. Εκρεμούν ακόμα κάποια τεχνικά ζητήματα στο θέμα αυτό. Είμαι πεπισμένος όμως ότι θα καταλήξουμε σε κάποια λύση. Όσον αφορά την κατάσταση εντός της Σλοβακίας, ε, αυτή είναι ο λόγος που βρίσκομαι εδώ σήμερα. Θα ήθελα να σας περιγράψω πώς βλέπουμε εμείς το Dieselgate. Καταρχάς, θα ήθελα να πω ότι όλα τα οχήματα που κατασκευάζονται στην Σλοβακία δεν λαμβάνουν έγκριση τύπου στην Σλοβακία. Αυτό συμβαίνει σε άλλες χώρες. Ε, στην κατηγορία μη δεν έχουμε εγκρίνει κανέναν τύπο. Τα περισσότερα οχήματα εγκρίνονται στην Γαλλία και κατόπιν στο Λουξεμβούργο και την Γερμανία και τις κάτω χώρες. μόνο τρέιλερ και τρακτέρ εγκρίνονται στη χώρα μας. Δηλαδή, κατηγορίες ε, που δεν ε, εμπίπτουν στο θέμα μας σήμερα. Η αρχή, η αρμόδια για την έγκριση τύπου στη χώρα μας ε, βρίσκεται στο Υπουργείο Μεταφορών, ε, ασχολείται όμως με άλλους τύπους οχημάτων όσον αφορά το Υπουργείο μας και την αρχή εποπτείας της αγοράς. Μετά από το ξέσπασμα του σκανδάλου αυτού, είχαμε σχετικές συζητήσεις και συναντηθήκαμε και με τους εκπροσώπους της Volkswagen. και η Σκότα, Audi και ΣΕΑΤ και Volkswagen μας υπέβαλαν προτάσεις για την λύση του θέματος που υποβλήθηκαν στο Υπουργείο για έγκριση. Όσον αφορά λοιπόν την βιομηχανία αυτοκινήτων, είμαστε μεγάλη αγορά Μπορώ να σας υποσχεθώ ότι η Σλοβακία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ε, λύσει το πρόβλημα αυτό που δημιούργησε το σκάνδαλο και ότι θα προσπαθήσουμε να βρούμε και λύση για το μέλλον. Τι έχει κάνει η Σλοβακία στο θέμα αυτό. Το θέμα των εκπομπών είναι σημαντικό για μας. Ε, ε, λαμβάνουμε μέτρα για την μείωση των εκπομπών. Θέλουμε να προωθήσουμε τις ε, σιδηροδρομικές μεταφορές. Ε, το 45% ε, της, του πληθυσμού της Σλοβακίας έχει δωρεάν μεταφορές στα τρένα. Και τα νέα οχήματα και μικρά αυτοκίνητα πληρώνουν χαμηλότερα τέλη από ό,τι τα παλαιότερα και μεγαλύτερα οχήματα. Επίσης, Έχουμε απλοποιήσει τους κανόνες ε, για τεχνικό έλεγχο των αυτοκινήτων. Ε, κυρίως μιλώ για τα παλαιότερα γιοταχή. Θέλουμε να ε, αποσύρουμε από τους δρόμους μας τα παλαιότερα και ρηπογόνα αυτοκίνητα. Δεν θέλουμε να γίνουμε νέο Detroit. Θέλουμε λοιπόν με τη βοήθεια νέων αυτοκινήτων ε, να δημιουργήσουμε ένα κλάστερ ε, για την κατασκευή οχημάτων. Είναι γνωστό ότι οι, κανόνες, οι ε, κινητήρες εσωτερικής καύσης δεν αποτελούν το μέλλον του τομέα αυτοκινήτων. Το μέλλον είναι τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα. Μείωση των εκπομπών ε, αποτελεί μέλλον της βιομηχανίας αυτοκινήτων. Άλλα μέτρα που υποστηρίζουμε είναι οι δοκιμές ε, και οι μετρήσεις εκπομπών υπό πραγματικές συνθήκες. Αυτό είναι ένα από τα θέματα της σημερινής συζήτησης. Ήδη υπόθηκε, ήδη ακούσαμε ότι έχει ολοκληρωθεί η έκθεση και εμφανίζομαι εδώ στην Επιτροπή σα μετά την ολοκλήρωση τη έκθεσης σε κάτι για το οποίο θα ήθελα να σας ζητήσω συγγνώμη. Είχαμε εκλογέ πέρσι. Τρεις διαφορετικού υπουργού είχαμε και είχαμε αναλάβει και την ε, Προεδρία ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία, αλλά παρακαλώ δεχτείτε τις ε, απολογίες μου που δεν μπόρεσα να παρευρεθώ νωρίτερα στην Επιτροπή σας. ανήκω στους υποστηρικτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, ο δρόμος δεν είναι εύκολος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά, είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι θα έχει περισσότερη επιτυχία στο μέλλον. Η Σλοβακία φυσικά εξαρτάται από την ζήτηση ε, για αυτοκίνητα στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζω η βιομηχανία αυτοκινήτων να μάθει από την σημερινή κατάσταση. Χρειαζόμαστε σαφέστερους κανόνες για το μέλλον. Σας ευχαριστώ και πάλι για την δυνατότητα να μιλήσω σήμερα εδώ στην Επιτροπή σας. Σας ευχαριστώ και την προσοχή σας. Είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε ερωτήσεις. Ευχαριστώ κύριε Στρόμτσεκ. Πρώτα οι εισηγητές, ο κύριος Κερμπράντη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον κύριο Στρόμτσεκ για την παρουσία του και την παρουσίασή του. Θα ήθελα να σας συγχαρώ και για την επιτυχή προεδρία σας. Ελπίζω να ξεκουραστήκατε τα Χριστούγεννα και να ανακτήσατε λίγο τον χαμένο ύπνο, διότι ξέρω ότι αυτό το εξάμεινο ήταν κουραστικό για σας. Το ερώτημά μου αφορά το Συμβούλιο, το Συμβούλιο ως θεσμικό όργανο. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος για τον οποίο είστε εδώ κατ' εμέ. Μιας και είχατε την Προεδρία εσείς ως Σλοβακία. Από το Σεπτέμβριο του 2015 <laughs> είδαμε ότι έγιναν πολλά. Το Κοινοβούλιο ξεκίνησε αυτήν την ε, ε Ερευνητική Επιτροπή, Εξαρτική Επιτροπή. Η Κομισιόν πολύ γρήγορα έκανε, υπέβαλε την αίτηση για την έγκριση τύπου. Ε, άνοιξαν διαδικασίες επί παραβάση από την Κομισιόν, αλλά το Συμβούλιο ως θεσμός σιώπησε. Έχω την εντύπωση ότι το μόνο που έκανε το Συμβούλιο ήταν να συζητά προτάσεις που προχώρησαν από την Κομισιόν. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι το εξής αφού του ξέσπασε το σκάνδαλο. Και ήταν πρωτοσέλιδο, παντού. Αφορούσε ένα βασικό δικαίωμα των πολιτών της Ευρώπης, ο καθαρός αέρας. Ε, γιατί δεν έγινε μια πραγματική συζήτηση πρώτο Συμβουλίου για το πώς συνέβη αυτό. Ως θεσμός, έτσι. Ξέρω ότι στα επιμερους κρατημέλη έγιναν συζητήσεις αλλά το Συμβούλιο είναι από τα βασικά θεσμικά όργανα, από τα τρία βασικά. Γιατί δεν έγινε η συζήτηση αυτή εκεί. Eh, σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Φυσικά, μπορώ να αναφερθώ σε αυτά που συνέβησαν ε, κατά το περασμένο εξάμεινο που είχαμε την Προεδρία. Η ισχύουσα οδηγία συζητήθηκε επί τέσσερα χρόνια μέχρι να καταλήξουμε σε κάποιο συμπέρασμα. Από τα 98 άρθρα τελικά ε, απομείνανε μόνο 50. 600 ε, σελίδες εκρεμούν ακόμα. Ε, που περιέχουν πολιτικές ερωτήσεις, πολιτικά θέματα. Τον Ιούλιο έγινε μια σχετική συζήτηση. Είμαι πεπισμένος ότι το πρόβλημα δεν προέκυψε το 2015 Ο καθένας από εμά που αγοράζει όχημα εξετάζει τον κατάλογο, εξετάζει τις τιμές που αναφέρονται και αναζητεί το όχημα με την βέλτιστη κατανάλωση. Ο καταναλωτής εξετάζει κυρίως το κόστος, ε, δεν εξετάζει τόσο πολύ την επιβάρυνση στο περιβάλλον. τα ε, τελευταία 20 χρόνια. Θα πρέπει να δούμε τι μέτρα πρέπει να ληφθούν ε, για να είναι συγκρίσιμες οι τιμές καταλόγου με τις πραγματικές τιμές. Εγώ αναφέρομαι στον πολιτικό ρόλο του Συμβουλίου ω θεσμικό όργανο. Πρόκειται για ένα ζήτημα που απασχολούσε του πολίτε. Το σύστημα, το σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ανταποκρίθηκε στο θέμα των εκπομπών του αυτοκινήτου. Ήταν τεράστια πολιτική κρίση. Όταν υπάρχει πολιτική κρίση, τότε άμεσα το θέμα εξετάζεται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ότι μιλάμε για τι πρόσφυγες, είτε για κάτι άλλο τέτοιου είδους κρίση ήταν και αυτή, σε έναν άλλο κλάδο, σε έναν άλλο τομέα. Αλλά στο Συμβούλιο επικράτησε σιωπή. Δεν συνέβη τίποτα. Πώς μπορεί κάποιος να ε, εμπιστευτεί το Συμβούλιο ως πολιτικό θεσμικό όργανο όταν σιωπή ε, προ μια τέτοιας κρίσης. Ε, Προσωπικά δεν πιστεύω ότι το Συμβούλιο σιωπά έχουν ε, ε, ληφθεί πολιτικά μέτρα και δεν νομίζω ότι να μα ενδιαφέρει μόνο αυτό που αναφέρεται στα μέσα μαζική ενημέρωση. πρέπει να μα ενδιαφέρουν τα πραγματικά αποτελέσματα, τα οποία μετά από έξι μήνε είναι σαφή. Έχουν διευκολυνθεί κάποιε διαδικασίε, έχουν επιταχυνθεί κάποιε διαδικασίε. αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν γίνει λάθη στο παρελθόν. Δεν είμαστε ρομπότ, άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε. Κανείς ε, δεν αμφισβητεί ότι έγιναν λάθη. Καταρχάς όμως ε, θα πρέπει να ασχοληθούμε με τα λάθη που έχουν γίνει. Είναι πολιτικό το πρόβλημα, μας ενδιαφέρουν οι πολιτικές παράμετροι. Ε, πρέπει να δημιουργήσουμε ένα τεχνικό πλαίσιο, κάτι που καταφέραμε κατά τη διάρκεια της Προεδρία μας ε, και Τώρα μπορούμε να ασχοληθούμε και με τα πολιτικά ζητήματα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριο Σκίζεκε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Υφυπουργέ που βρίσκεστε εδώ σήμερα στην Επιτροπή μας ε, μετά από την ε, δύσκολη για σας Προεδρία. Ε, στην εισαγωγή σας είπατε ότι είσαστε πρωταθλητές ε, στην ε, κατασκευή αυτοκινήτων. Συγχαρητήρια, το 2015 κατασκευάσατε πάνω από ένα εκατομμύριο οχήματα. Κατέχετε το παγκόσμιο ρεκόρ όσον αφορά την κατασκευή αυτοκινήτων ανακάτοικο. Τα αυτοκίνητα που κατασκευάζονται, πόσα από αυτά είναι διζελοκίνητα. Πρέπει να ομολογήσω ότι δεν έχω τον ακριβή αριθμό. Νομίζω όμως ότι ακολουθούμε τον μέσο όρο της Ευρώπης. Ε, τα περισσότερα αυτοκίνητα που κατασκευάζονται στην Ευρώπη εξάγονται. Ε, αν λοιπόν εξετάσουμε το ποσοστό διζελοκίνητων ε, αυτοκινήτων στην Ευρώπη, νομίζω ότι στην Σλοβακία έχουμε αντίστοιχο αριθμό ο κύριος Κίζικε. Αρχικά είπατε ότι έχετε αρκετά μεγάλο ποσοστό διζελοκίνητων αυτοκινήτων, πάνω από 50%. Και αυτό οφείλεται και σε αυτά που υπογορεύει η πολιτική για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, μπορείτε να μας το διευκρινίσετε αυτό. Μήπως θα μπορούσατε να ε, συγκεκριμενοποιήσετε την ερώτησή σας. Ανέφερα ότι στο παρελθόν ασκήθηκε πίεση από πλευρά των καταναλωτών διότι αναζητούσαν κυρίως σε χαμηλό κόστος. Τα διζελοκίνητα είχαν χαμηλότερη κατανάλωση, το δίζελ ήταν και πιο φτηνό από τη βενζίνη και Γι' αυτό στο παρελθόν είχαμε πολλά διζελοκίνητα αυτοκίνητα. Σήμερα αλλάζει αυτό. Οι κατασκευαστές οχημάτων ε, προσανατολίζονται περισσότερο στα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα, καθώς ε, και σε εναλλακτικά καύσιμα. «46.000 οχήματα καταχωρήθηκαν ε, στο, στην Σλοβακία» ο κύριος Γκίζε και ασχολούμαστε με την έγκριση τύπου και οι εργασίες της Επιτροπής μας θα αποτελέσουν και υπόδειγμα για την ε, η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς. Κατά την εισαγωγή σας είπατε ότι αναέτος ε, παράγεται ένα εκατομμύριο οχήματα ε, στην Σλοβακία, αλλά έγκριση τύπου πραγματοποιείται μόνο για τα τρέιλερ και για τα τροχόσπιτα. Ε, η έγκριση τύπου γίνεται στη Γαλλία, στο Λουξεμβούργο. Στην Ευρώπη πάντα μας ε, μιλάνε για την Επιτροπή της Επικουρικότητας, κάτι που μπορεί να λυθεί επιτόπου, να λυθεί επιτόπου. με τις εμπειρίες σας από το Υπουργείο Μεταφορών προτείνετε μεταρρύθμιση της έγκρισης τύπου και της εποπτείας της αγοράς. Ε, πώς έχουν τα πράγματα στη χώρα σας. Από τη μία, συζητήσαμε σήμερα το πρωί ότι ζητείτε περισσότερη Ευρώπη, κεντρική ε, ρύθμιση δηλαδή. Κάτι που μπορεί να περιορίσει τα δικαιώματα των κρατών μελών. Από την άλλη θα πρέπει να γίνεται η έγκριση εκεί όπου κατασκευάζονται τα, τα αυτοκίνητα. Ε, εσείς ε, πώς βλέπετε την κατάσταση αυτή. Κατάλαβα την ερώτησή σας. Η Σλοβακία ακολουθεί το σύστημα που έχει εισάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχουμε εμεί τη δυνατότητα να πούμε πού θα πρέπει να γίνονται οι δοκιμές. Ο κατασκευαστής διασφαλίζει την ασφάλεια και οι εκπομπές αποτελούν μόνο ένα μέρος της ε, συνολικής έγκρισης. Θα θέλαμε να ενισχυθεί η θέση της Ευρώπης κατά τους ελέγχους και κατά την εποπτεία. Εμείς δεν έχουμε αντίρρηση τα οχήματα να ε, εγκρίνονται στη χώρα όπου κατασκευάζονται. Από την άλλη έχουμε ενιαία εσωτερική αγορά ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και η αρχή του ελέγχου στην χώρα κατασκευής ε, αντίκειται στις αρχές της ενιαίας αγοράς. Όταν κατασκευάζεται ένα προϊόν σε μια χώρα θα πρέπει να μπορεί να κυκλοφορήσει στο σύνολο της Ευρώπης. Αμοιβαία αναγνώριση δηλαδή της έγκρισης τύπου. Συνοψίζοντας να πω ότι αποδείχθηκε ότι το σύστημα του παρελθόντος δεν ήταν καλό. Και με το νέο κύκλο δοκιμών ε, έχουμε επιτάχυνση της διαδικασίας. Αυτό είναι θετικό και θα είναι θετικό να εισάγουμε μια κεντρική διαδικασία. Στις Βρυξέλλες γίνονται τέτοιες συζητήσεις. Οι πρώτες συζητήσεις δείχνουν όμως ότι κάτι τέτοιο θα είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Η Σλοβακία σίγουρα δεν μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφορά για το σύνολο τη Ευρώπη. Εμεί είχαμε προβλήματα κατά του τεχνικού ελέγχου οχημάτων στη χώρα μα. τροποποιήσαμε την νομοθεσία και τώρα πια έχουμε μηδενική ανοχή. Σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι κανόνες, ε, αφαιρούνται οι άδειε και δεν μπορεί να παρακάμψει κανείς τους κανόνες για να παρουσιάζει καλύτερη εικόνα απέναντι στους καταναλωτές. Αυτό δεν συμφέρει πια τους ε, κατασκευαστές αυτοκινήτων. Παρομοίως, κατά την έγκριση τύπου ε, των οχημάτων ε, μπορεί να γίνει κάτι ανάλογο. ώστε να λαμβάνονται μέτρα σε περίπτωση που οι αρχές δεν πληρούν τις υποχρεώσεις τους. Να υπάρχει δηλαδή μια αλυσίδα ευθύνης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό εξηγεί και την ε, απάντησή σας στην ερώτηση 1, όπου αναφερθήκατε στην ε, δημιουργία επιπλέον γραφειοκρατίας. Λέτε όμως ότι θέλετε και περισσότερη ε, ευρωπαϊκή αρμοδιότητα. Και μία τελευταία ερώτηση σχετικά με την εισαγωγή σας. Μιλήσατε πολύ αρνητικά όσον αφορά το μέλλον ε, του κινητήρα εσωτερικής καύσης. Εύκολα μιλάει κανείς για το μέλλον της ηλεκτροκινητικότητας. Εγώ θέτω εδώ μεγάλο ερωτηματικό, διότι η ηλεκτροκινητικότητα θα είναι βιώσιμη μόνο ε, εφόσον ε, και το ηλεκτρικό ρεύμα παράγεται με τρόπο βιώσιμο. Ε, αν δηλαδή έχουμε θερμοελεκτρικό εργοστάσιο με, με λιγνίτη, τότε δεν θα έχουμε βιώσιμη ηλεκτροκινητικότητα. Ίσως θα πρέπει λοιπόν να ακολουθήσουμε διτή οδό στο μέλλον, διτή προσέγγιση. Φυσικά χρειαζόμαστε δίτη προσέγγιση, όπως πολύ σωστά είπατε. Πρέπει να βελτιώσουμε την κατάσταση ήδη σήμερα. Δεν αποτελεί λύση το να πούμε ότι είναι προβληματικοί οι σημερινοί κινητήρες και το μέλλον ανήκει αποκλειστικά στα εναλλακτικά καύσιμα. Θα πρέπει να εξετάσουμε τη σημερινή κατάσταση. Πολλοί κινητήρες ε, δημιουργούν πολλούς ρήπους. Χρειαζόμαστε όμως οχήματα για τη δουλειά μας. Ε, δεν μπορούμε ε, να τα καταργήσουμε τελείως. Γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται ρητή προσέγγιση. Στην Σλοβακία προτιμάμε τα γιοταχή που ρηπαίνουν λιγότερο το περιβάλλον. καθώς και οχήματα με μικρότερο κυβισμό. Είναι πιο εύκολη η καταχώρησή τους και είναι χαμηλότερα τα τέλη για τα οχήματα χαμηλότερου κυβισμού. Προσπαθούμε επίσης να επηρεάσουμε την συμπεριφορά των ε, οδηγών ώστε να ε, λαμβάνουν αποφάσεις πιο φιλικές προς το περιβάλλον. Σε κεντρικό επίπεδο πρέπει να το συζητήσουμε αυτό. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στο παρελθόν, στη Φόρμουλα 1 ε, επιτρεπόταν να χρησιμοποιεί κανείς κινητήρες που μπορούσε να την καταστήσει κανείς μετά από κάθε αγώνα μιας χρήσης. Μετά όμως δημιουργήθηκαν κανόνες ώστε να μπορούν να συμμετέχουν ε, και άνθρωποι που δεν ε, έχουν ε, οικονομική, δυνατότητα να αλλάζουν τον κινητήρα κάθε φορά. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε τι κινητήρες εγκρίνουμε για την καθημερινή μετακίνηση. Θα μπορούσαμε να κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα σε ρηπογόνα και λιγότερα ρηπογόνα αυτοκίνητα ε, στους δρόμους. Είμαι πεπισμένος ότι το μέλλον ανήκει στις εναλλακτικές μορφές ε, μετακίνησης, ε, όχι στους κινητήρες εσωτερικής καύσης και τους διζελοκινητήρες. Θα πρέπει όμως να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να μειώσουμε τους ρήπους. Τα ηλεκτροκίνητα, αυτοκίνητα λοιπόν είναι το πιο σημαντικό στοιχείο εδώ και θα πρέπει φυσικά, συμφωνώ μαζί σας, ε, να επιφέρουμε αλλαγές ε, και στην ε, παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, να μην έχουμε δηλαδή ε, εργοστάσια θερμοελεκτρικά με λιγνίτη. Θα δούμε σημαντικές αλλαγέ και κατά την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος και στην κατασκευή οχημάτων στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κριστίν Λοβού έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ που ήρθατε στην Επιτροπή, την Εξεταστική. Ίσως θα ήταν πιο σημαντικό να μπορούσαμε να σας δεχτούμε στην ακρόαση όταν δεν είχαμε τελειώσει την ακρόαση, κυρίως όταν συλλέγαμε όλα τα στοιχεία. Και δεν μπορούμε να συμπεριλάβουμε αυτά που συζητούμε σήμερα, διότι ολοκληρώθηκε η έκθεση του του λεχθέντος. Εξετίμησα το ότι είπατε ότι θα έπρεπε να δοθεί ευρωπαϊκή απάντηση στην όλη κατάσταση. Μια γενική απάντηση χρειάζεται, συστημική απάντηση είναι κάτι με το οποίο συμφωνούμε μαζί σας. Πάνω σε αυτό θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η απόψή σας. Θα ήθελα μια απάντηση όσον αφορά το σύστημα για το σεβασμό της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας σε όλη την κλίμακα κατασκευής. Τι σκεφτόσαστε για μια ανεξάρτητη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία η οποία θα μπορούσε να εποπτεύει σε περίπτωση που οι εθνικές αρχές που δίνουν την έκκληση τύπου των οχημάτων ε, θα είχαν κάποια προβλήματα. Θα μπορούσε να είναι μια λύση. Είναι μια επιλογή που προτείνουμε και συζητούμε. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό. Σαν Σλοβάκος Υπουργός, σαν Υπουργός σαν σκάτους μέλους, ποια είναι η άποψή σας και ως Προεδρεύων του Συμβουλίου επί ένα εξάμεινο. Ποια είναι η άποψή σας επ' αυτού. Ε, σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ σύντομη απάντηση. Ναι. Πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι Βρυξέλλες γενικότερα θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερες αρμοδιότητες από ό,τι στο παρελθόν. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ε, ένα κατάλληλο μέσο. Θα μπορούσε ο οργανισμός αυτός να είναι ένα κοινό κέντρο ερευνών. Ήδη ανέφερα ότι μπορεί να παίζει ρόλο ελεγκτή. Να εξετάζει αν ε, τηρούνται όλοι οι κανόνες και εάν τα οχήματα συμμορφώνονται με τους κανόνες. Αυτή η κοινή αρχή θα μπορούσε να διενεργεί Έχουμε το ε, κοινό αυτό Συμβούλιο Ερευνών, το GRC. Ε, ποτέ όμως δεν είχε εντολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτός ο φορέας για να εξετάζει αν όλα γίνονται σωστά. Είναι κάτι που πρέπει να διορθώσουμε. Δεύτερη ερώτηση αφορά την απάντηση που δώσατε στην ερώτηση 5 και που αναφέρατε στην ομιλία σας. Τους επιθεωρητές σας που έκαναν έρευνες στους κατασκευαστές αυτοκινήτων. Μπορείτε να πείτε περισσότερα για τα απορίσματα των ερευνών τους. Ζητήσατε αυτοί οι επιθεωρητές να ελέγξουν αν υπήρχαν μηχανισμοί αναστολής. Βρέθηκαν. Αν είχατε αποτελέσματα, τι κάνατε διότι αναφερθήκατε στη Volkswagen που παράγει αυτοκίνητα στη χώρα σας. Να διορθώσω, κανένα όχημα που κατασκευάστηκε στη Σλοβακία δεν έλαβε έγκριση τύπου στη Σλοβακία. Όλες οι συζητήσεις μας με μεμονωμένους κατασκευαστές έγιναν για να μάθουμε τη θέση των κατασκευαστών. Στις συζητήσεις μας ε, ήταν σημαντικό να γνωρίζουμε πώς μπορεί να αφαιρεθεί το λογισμικό που έχει τοποθετηθεί αντίθετα με τους κανόνες. 36 μοντέλα Volkswagen, Audi, Skoda και Seat αφορούσε αυτό το θέμα. Μιλήσαμε λοιπόν για την αφαίρεση του λογισμικού και γίνονται επιχειρήσεις αντικατάστασης τους. Ε, η τελευταία τέτοια έγινε τον Δεκέμβριο του 2016. Ο έλεγχος των οχημάτων όμως ε, απαιτεί τροποποίηση του συστήματος. Ε, η Σλοβακία στο μέλλον θα ασχοληθεί με την αλλαγή του συστήματος αυτού, διότι όπως υπόθηκε δεν θέλουμε να συνδεθούμε με τις ε, απατηλές πρακτικές των κατασκευαστών. Θέλουμε οι τιμές που αναφέρονται στον κατάλογο των αυτοκινήτων να είναι και οι πραγματικές. Θέλουμε λοιπόν αυτοκίνητα με χαμηλέ εκπομπέ και ε, με υψηλά πρότυπα ασφαλεία για το σύνολο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριος Χερμπράντη, πρόεδρε, θα ήθελα να επανέλθω σε κάτι που ο κύριος Τρόμτσεκ ανέφερε. Στον πρώτο γύρο ερωτήσεων απαντήσεων. ότι συζητούμε τεχνική φύσεω πρόβλημα και όχι πολιτική φύσεω, είπε. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι το σωστό συμπέρασμα. Έχουμε αρκετά ισχυρά συμπεράσματα στην έκθεσή μα. Εκεί λέμε ότι λόγω πολιτικών αποφάσεων δημιουργήσαμε το πρόβλημα το οποίο κατέληξε να γίνει Dieselgate. Για μία ακόμη φορά λοιπόν θέτω το ερώτημα αυτό είναι ένα τεράστιο πολιτικό πρόβλημα. Είδαμε ότι το ευρωπαϊκό σύστημα δεν λειτουργεί καλά. Είδαμε ότι τα κράτη-μέλη δεν εφαρμόζουν τους ευρωπαϊκούς κανόνες σωστά. Ότι κάποιοι πολιτικοί έλαβαν πολιτικές αποφάσεις εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ούτω ώστε να παρακάμψουν, να παρεμποδίσουν το σύστημα που δημιουργήσαμε. Και το κόστος ε, είναι ότι όλα αυτά έγιναν εις βάρος 500 εκατομμυρίων ε, πολιτών, Ευρωπαίων πολιτών που δεν έχουν καθαρή ατμόσφαιρα όπως θα έπρεπε. Για μία ακόμη φορά ρωτώ, γιατί το Συμβούλιο σαν θεσμό, σαν θεσμικό όργανο δεν έκανε τίποτα με την πολιτική κρίση που κρύβεται πίσω από το Dieselgate και αυτό είναι εντελώς διαφορετικό από τη συνθισμένη διαδικασία που ήδη εφαρμοζόταν για το RDE, εγκρίσεις τύπου κλπ. Αυτό είναι κάτι άλλο. Δεν αντιμετωπίζει τις πολιτικές κρίσεις με αυτόν τον τρόπο ένα ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο όπως το Συμβούλιο. Εξηγήστε μου, σαν θεσμός το Συμβούλιο, σαν το μόνο ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο που δεν κάνει τίποτα, αποφάσισε να μην κάνει κάτι. Προσωπικά, δεν θεωρώ ότι το Συμβούλιο δεν έχει κάνει τίποτα. Επαναλαμβάνω τη θέση μας. Συμφωνώ μαζί σας ότι πρόκειται για πολιτικό πρόβλημα. Είναι κάτι που αφορά πάρα πολλούς καταναλωτές, σχεδόν τον καθένα. Ε, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά είναι πολιτικό ζήτημα, φυσικά είναι πολύ ευαίσθητο ζήτημα. Δεν διαφωνώ. Αλλά φυσικά έχει προκληθεί το ε, θέμα αυτό από λυπή τεχνικά πρότυπα. Το τεχνικό σύστημα απέτυχε. Καταρχάς λοιπόν θέλαμε να λύσουμε τα, τις τεχνικές εκκρεμότητες και κατόπιν, όπως είπα και στην εισαγωγή μου, να συζητήσουμε από κοινού τα εκρεμή πολιτικά ζητήματα. Συζητάμε λοιπόν ε, το θέμα εάν θέλουμε οργανισμό ή όχι, ποιες ε, πρέπει να είναι οι αρμοδιότητες ε, των κρατών μελών, εάν θέλουμε να περιορίσουμε τις αρμοδιότητες των κρατών μελών ή όχι. Όλα αυτά θα πρέπει να τα συζητήσουμε ανοιχτά. Η Σλοβακία δεν έχει πρόβλημα με μια λύση που θα οδηγήσει σε καλύτερη συστημική λύση και που θα αποτρέψει παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον. Το σύνολο της δομής εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, αλλάζει. Ασχολούμαστε όμως με το θέμα και γι' αυτό πετυχαίνουμε καλύτερα αποτελέσματα. Άλλο θετικό παράδειγμα που θα ήθελα να αναφέρω ε, στον τομέα της επικοινωνίας είναι η πρόταση για τα τέλη περιαγωγής. Επί χρόνια ο καθένας υπολόγιζε διαφορετικά τα τέλη περιαγωγής. Ε, τώρα πια, χάρη στην απόφαση των Βρυξελών, έχουμε μια συστημική λύση οικονομική και φιλική προς τον πελάτη. Μπορώ να σας αναφέρω και άλλα τέτοια θέματα που δείχνουν ότι είχαμε θετικά αποτελέσματα από τις Βρυξέλλες. Είμαι πεπισμένος ότι ετούτη η περίπτωση αποτελεί αντίστοιχη ευκαιρία. Θα απαιτηθεί αρκετός χρόνος και αναφέρθηκα στην περίπτωση όπου ο πελάτης βλέπει άλλες τιμές στον κατάλογο. Θα πρέπει λοιπόν όμως όπως είπα πρώτα να ρυθμίσουμε τα τεχνικά ζητήματα και κατόπιν να ακολουθήσει η πολιτική συζήτηση η οποία πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή και κατόπιν να κλείσουμε το θέμα. Δεν θα ήταν σωστό πρώτα να ασχοληθούμε με τα πολιτικά συμπεράσματα. Πρώτα θα πρέπει να γίνουν οι τεχνικές ρυθμίσεις, να δούμε τι θα πρέπει να αλλάξει. και θα χρειαστούμε αργότερα πολιτική συμφωνία. Ευχαριστώ κυρία Κονέσκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω και τον Υπουργό που ήρθε για την ακρόαση για να μας εξηγήσει τις θέσεις της Σλοβακίας Αντιλαμβάνομαι τη θέση σας σε ό,τι αφορά τη σημασία της αυτοκρατοβιομηχανίας, το καταλαβαίνω και ως ε, ε Τσέχα και εμείς ε, σε μια παρεφερή <coughs> θέση είμαστε σε ό,τι αφορά το τι αντιπροσωπεύει το κοινοβιομηχανία σε επίπεδο ΑΕΠ, σε επίπεδο απασχόλησης και πόσο ευαίσθητος είναι αυτός ο κλάδος για την οικονομία μας και κρίσιμος. Καλό θα ήταν να μιλήσουμε και για το παρελθόν όμως, όχι μόνο για το μέλλον. Εδώ κάποιος κοράδεψε τους καταναλωτέ Και οι Ευρωπαίοι καταναλωτές ε, θα πληρώσουν πολύ περισσότερο από τις ΗΠΑ ή ε, στην Νότια Κορέα όπου αυτή τη στιγμή έχουν ξεκινήσει διαδικασίες ε, και οι καταναλωτές αποζημιώνονται ενώ οι, οι χιλιάδες, οι εκατοντάδες χιλιάδες αγοραστές αυτοκινήτων που καλόπιστα αγόρασαν αυτά τα οχήματα δεν μπορούν να προστατεύσουν τον εαυτό τους τη στιγμή. Πώς πιστεύετε πρέπει να το, να αυτό. Θα πρέπει να, για να κλείσουμε το θέμα, να εξηγήσουμε στους Ευρωπαίους καταναλωτές πώς θα τους προστατεύσουμε στο μέλλον. Αλλά πρέπει να δούμε και τι θα γίνει με αυτούς που ζημιώθηκαν τώρα που ήταν θύματα αυτής της απάτης τώρα που αγόρασαν αυτά τα αυτοκίνητα διότι θέλουν να μειώσουν τις εκπομπές τους. Τι θα γίνει με αυτό. Καταρχάς, θα ήθελα να πω ότι εκρεμούν κάποιες δικαστικές υποθέσεις. Η καταναλωτές έχουν πάντα τη δυνατότητα να ε, προσφύγουν στα δικαστήρια. Κατά τη γνώμη μας είναι πιο σημαντικό να δημιουργήσουμε καλούς κανόνες για το μέλλον. Δεν μπορούμε να διορθώσουμε το παρελθόν. θα μπορούσα να σας ρωτήσω και εσάς ε, τι έγινε στο παρελθόν για να αποτραπεί το σκάνδαλο. Είναι σημαντικό όμως να βγάλουμε τα κατάλληλα συμπεράσματα και να αποφύγουμε τέτοιες καταστάσεις στο μέλλον. Ένας οδηγός όταν σκέφτεται την αγορά νέου αυτοκινήτου δεν θα πρέπει να επηρεάζεται υπερβολικά από το σκάνδαλο Dieselgate. Ο καταναλωτής εξετάζει το κόστος, την ασφάλεια κλπ. και αναζητεί κατάλληλο μοντέλο συγκεκριμένης κατηγορίας. Δεν μπορούμε να υπολογίσουμε την αντίδραση του καταναλωτή στο σκάνδαλο αυτό. Σημαντικό για μας είναι το τι κάνουμε εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι το τι γίνεται στις Ηνωμένε Πολιτείες. Πρέπει να ασχοληθούμε με το τι γίνεται στις χώρες μας και να ευχηθούμε ε, όλα τα καλά στους ε, γειτόνους μας. Όσοι ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν δικαίωμα να εισπνέουν καθαρό αέρα. Και έχουν ε, επίσης το δικαίωμα να αγοράζουν ε, ε, αξιόπιστα αυτοκίνητα με προδιαγραφές που να αντιστοιχούν σε αυτές που υπάρχουν στον κατάλογο. Εάν το πετύχουμε αυτό, νομίζω ότι αυτό θα είναι καλή έκβαση του σκανδάλου αυτού. Όσον αφορά τις δικαστικές προσφυγές ε, μεμονωμένων καταναλωτών, δεν είμαι εμπειρογνώμων, αλλά νομίζω ότι στην ομοθεσία αναφέρεται κάτι σχετικό, στην οδηγία αναφέρεται. Όταν λέτε το πώς πρέπει να συναγάγουμε μαθήματα και είπατε πώς αντιμετωπίσετε το θέμα στο Συμβούλιο και κατά πόσο θέλουμε μια νέα ευρωπαϊκή υπηρεσία η οποία θα ελέγχει και θα εποπτεύει, το αναφέρατε αυτό, μιλήσατε όμως για το ποιες διαδικασίες θα πρέπει να θεσπιστούν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής ώστε να μην επαναληφθεί το φαινόμενο. Διότι είναι σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνώριζε αρκετά χρόνια πριν ότι υπήρχαν αυτοί οι μηχανισμοί αναστολής και χρησιμοποιούνται. Είχαν πληροφορηθεί από διάφορες πηγές, αλλά ποτέ δεν έκαναν τίποτα. Δεν έλαβαν μέτρα μέχρι ότου τελικά φανερώθηκε αυτό στα μέσα ενημέρωσης και δημιουργήθηκε ένα πολιτικό σκάνδαλο. Μιλήσατε σε επίπεδο Συμβουλίου πώς θα αντιμετωπιστούν οι διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πώς θα βελτιωθούν οι διαδικασίες που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι αυτό είναι πρόβλημα που θα πρέπει να απευθύνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν μπορώ να μιλήσω εδώ στο όνομά της. Παρ' όλα αυτά, εγώ είμαι πεπισμένος ότι θετικό στοιχείο Ε, είναι ότι μειώνεται όλο ένα και περισσότερο η ανοχή των πολιτών. Στη Σλοβακία, για παράδειγμα, δεν γίνεται πια αποδεκτή η σιωπή σε περίπτωση ε, κάποιου ερωτήματος. Ε, τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης έχουν οδηγήσει σε τέτοια αρνητική ανοχή. Συχνά αναφέρεται κανείς με αρνητικό τρόπο σε αυτά, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ε, αλλά βλέπουμε όλο και πιο γρήγορες αντιδράσεις. Ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μάθει από αυτό και να προσεγγίσει με καλύτερο τρόπο τα προβλήματα. Να επανεξετάσει τις δικές της ε, διαδικασίες. Θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε καλύτερες διαδικασίες στο μέλλον. Δεν μπορούμε να αγνοούμε τις ε, παρατηρήσεις και τα μηνύματα των πολιτών. Ελπίζω στο μέλλον να σημειώσουμε πρόοδο στο θέμα αυτό. Ο κύριος Σέκχαρτ, να το Ευχαριστώ, ευχαριστώ κυρία Στρόμψεκ, ε, τον κύριο Στρόμψεκ μάλλον για την εισαγωγή του και τις απαντήσεις του. Όπως ε, θα διαπιστώσατε, ε, εδώ όλοι λέμε ότι το σκάνδαλο είναι τεράστιο και αυτό είναι λυπηρό για την Ευρώπη και αυτό που μας ενοχλεί να εξετάζουμε το επίπεδο της λήψης από των αποφάσεων ακόμα και μετά το ξέφυγμα του σκανδάλου δεν φαίνεται να επίγεστε να το αντιμετωπίσετε. Λέτε ότι είχατε κάποιες συζητήσεις, ναι, αλλά να σας πω και κάποιες θέσεις, έτσι, που ακόμα παίρνει η Σλοβακία μετά το σκάνδαλο, του Dieselgate. Η συζήτηση για το RDE, το δεύτερο πακέτο, για, τις, ε, για τη συμμόρφωση. Θέλετε πέντε χρόνια καθυστέρηση στην εφαρμογή σε σχέση με την πρόταση της Κομισιόν, έτσι. Ζητάτε να αργήσει να καθυστερήσει πέντε χρόνια. Ακόμα και για το τεστ RDE, έτσι, που είναι τόσο κρίσιμο. Πραγματικά δυσκολεύομαι ιδιαίτερα να το καταλάβω αυτό, ενώ την άλλη λέτε ότι επήγει το θέμα. Και το άλλο, για τη συμμόρφωση. Η Σλοβακία λέει ότι από τη στιγμή που το RD χρησιμοποιείται για τη συμμόρφωση δεν πρέπει να υπάρχει δυνατότητα κάποιος νομοθέτης αργότερα ή κάποιος τρίτος να δοκιμάσει εκ νέου ε, με RDE κατά πόσο αυτός ο παράγοντας ε, συμμόρφωσης ε, ισχύει. Είστε κατά δηλαδή αυτής της δυνατότητας. Και αυτό είναι εξαιρετικά περίεργο. Όταν ξέρουμε ότι είναι λίγη έλεγχη. Γιατί παίρνει αυτές τις θέσεις η Σλοβακία. Ε, Θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Εγώ δεν έχω ακούσει να απορρίπτουμε νέους ελέγχους. Πάντα λέγαμε ότι χρειαζόμαστε συστημικές λύσεις και όσον αφορά το πρώτο μέρος ε, της ερώτησής σας. Θέλαμε ενιαίους κανόνες ε, για όλους τους ε, τύπους και γι' αυτό έχουμε απόσχει από την ψηφοφορία. Όταν δημιουργείται ένα νέο όχημα στην βιομηχανία αυτοκινήτων, Ο σχεδιασμός απαιτεί πολύ χρόνο προτού να καταλήξει το όχημα στο δρόμο. Και η έγκριση απαιτεί χρόνο. Απαιτείται πολλή δουλειά κατά το σχεδιασμό ενός ε, οχήματος ε, για τον κινητήρα και για άλλα θέματα. Χρειάζεται λοιπόν ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα. Επίσης, σε ένα ποδήλατο είναι πολύ εύκολο να αλλάξει κανείς αλυσίδα, αλλά στην ε, βιομηχανία αυτοκινήτων ο σχεδιασμός ενός νέου αυτοκινήτου και η έγκρισή του απαιτούν πολύ χρόνο. Δεν είμαστε κατά των δοκιμών RDE, όπως λέτε εσείς, απλά θέλουμε σαφείς και ενιαίους κανόνες, ρεαλιστικούς που να μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη. On the first point, on the of, uh, uh, Για το πρώτο που είπατε ε, για τη συμμόρφωση, ε, κοιτάξτε στα πρακτικά ποια είναι η θέση σας. Ε, Τώρα για την καθυστέρηση 5 ετών στην οποία αναφερθήκατε. Αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ Πολιτείες αυτές οι ίδιες μάρκες έχουν αυτοκίνητα με νέες τεχνολογίες που τίθεται ήδη προς πώληση στην αγορά. Μπορούν να το κάνουν λοιπόν οι μηχανίες αλλά δεν το κάνουν στην Ευρώπη γιατί ξέρουν ότι η έλεγχη δεν είναι τόσο αυστηρή. Και ερχόμαστε σε άλλο, μια άλλη θέση τώρα της Σλοβακίας. Σε ό,τι αφορά την συμμόρφωση ε, την υπηρεσιακή, λέτε ότι μόνο ε, το bench πρέπει να ελέγχεται. Και αυτό είναι εξαιρετικά περίεργο. Γιατί... Skúsim najprv zareagovať na tú kontrolu, ktorú ste porovnali s Amerikou. A tu je tá θα προσπαθήσω να απαντήσω στη σύγκρισή σας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω ότι εδώ έχουμε μια ιδιαίτερη ευκαιρία για τις Βρυξέλλες. Εγώ αν ήμουν κατασκευαστής θα έκανα μόνο τα απολύτως απαραίτητα. Στόχος μου είναι να κερδίσω χρήματα. και οι κατασκευαστές προσπάθησαν να κερδίσουν όσο περισσότερα χρήματα από τον καταναλωτή πριν την παρέμβαση των Βρυξελών. Οι κατασκευαστές θέλουν οικονομικά αποτελέσματα. Οι Βρυξέλλες λοιπόν έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν κεντρικό φορέα ελέγχου. Και όσον αφορά το δεύτερο τμήμα της ερώτησής σας, ήδη κατά την εισαγωγή μου, ανέφερα ότι οι έλεγχοι υπό πραγματικές συνθήκες οδήγησης αποτελούν ε, την μόνη δυνατότητα για το μέλλον. Ποτέ δεν ήμασταν κατά αυτού. Αλλά απαιτήσαμε ίδιες προθεσμίες ε, για όλα τα ίδια ελέγχων. Θα με ενδιαφέρε πολύ να μάθω πότε η Σλοβακία ισχυρίστηκε αυτό που λέτε. Οι συνάδελφοί μου συμμετέχουν σε κάθε συνεδρίαση και δεν έχουν λάβει τις πληροφορίες που μου αναφέρατε. Ίσως θα μπορούσαμε διμερώς να το συζητήσουμε μετά το τέλος της σημερινής συνεδρίασης. Ευχαριστώ. Πάμε στο δεύτερο γύρο των ερωτήσεων. Τρία λεπτά στον καθένα. Ο κ. Βάντερ Κάμπ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό που ήρθε. Τον ευχαριστώ και για τις απαντήσεις του. Εν γέννη απαντήσεις του υπήρξαν σαφείς στην εισαγωγή σας. Είπατε κάτι ενδιαφέρον που αφορούσε τα είδη των αυτοκινήτων που παράγεται. και ότι η έγκριση τύπου χορηγείται σε άλλες χώρες. Ποια είναι η εμπειρία σας από αυτό το σύστημα. Το θεωρείτε κάτι αποδεκτό ή αισθάνεστε ότι θα προτιμούσατε οι αρχές της Σλοβακίας να εμπλέκονται στη διαδικασία αυτή. Μου λέτε ε, ότι άλλοι κάνουν τη, δίνουν την έγκριση τύπου και εσείς παράγετε αυτοκίνητα. Ε, εσύ, ποια είναι η άποψή σας, θα προτιμούσατε να είναι διαφορετικά τα πράγματα. το ako som hovoril, sme súčasťou Γενικά, να πω ότι ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και χαιρόμαστε που ισχύει η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας ε, και ελεύθερης διακίνησης ε, αγαθών. Είμαστε χώρα που επικροτεί τους ενιαίους φορείς, τα, κοινο... τα κοινά κέντρα ελέγχου και ερευνών. Από την άλλη, Εάν έχουν εγκριθεί οχήματα σε κάποιο μέρος ε, της Ευρώπης, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα το να γνωρίσουμε, εφόσον έχουν ε, τηρηθεί οι προδιαγραφές, εφόσον οι δοκιμές αυτές έχουν γίνει με σωστό τρόπο. Σε περίπτωση λοιπόν που δούμε αλλαγές και που ε, τα οχήματα πρέπει να ε, ε, ελέγχονται, να περνούν δοκιμές στην χώρα κατασκευής, δεν έχουμε πρόβλημα με κάτι τέτοιο. Ούτε έχουμε πρόβλημα να αναγνωρίσουμε οχήματα που έχουν εξεταστεί σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημαντικό για μας είναι μαζί με τις Βρυξέλλες να δημιουργήσουμε ένα σύστημα που να αποτρέπει τις αθέμητες πρακτικές. Είναι σημαντικό για ε, ε, η διαδικασία έγκρισης ε, να πραγματοποιείται με τρόπο σωστό. Ευχαριστώ. Η δεύτερη ερώτησή μου αφορά αυτή την υπηρεσία στο Κοινοβούλιο. Έγιναν διάφορες συζητήσει, έντονες συζητήσει όσον αφορά τα υπέρ και τα κατά ενό φορέα, αν θα ήταν καλύτερα τα πράγματα αν είχαμε κάποιον τέτοιο φορέα. Είπατε ότι η πλευρά Σλοβακία θα θέλατε να υπάρχει ένα φορέα. Μπορείτε να το ξεκαθαρίσετε αυτό. Γιατί θέλετε να υπάρχει ένας τέτοιος φορέας. Άλλη ερώτηση σχετική. Πώς ε, προς τα πού οδεύουν οι συζητήσεις από αυτού στο Συμβούλιο σε αυτή τη φάση. Spojím obidve otázky do jednej, lebo myslím θα απαντήσω από κοινού στις ερωτήσεις αυτές. Πιστεύουμε ότι πρέπει να αλλάξει το σύστημα. Και πρέπει να αποφύγουμε νέα σκάνδαλα. Το πώς θα λειτουργεί ο σχετικός οργανισμός ε, θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο πολιτικής συζήτησης. θα πρέπει πολιτικά να συζητηθεί το πώς ε, μπορούν να παρέμβουν τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να υπάρχει εποπτεία όλων ε, των ελέγχων και στα κράτη-μέλη. Δεν είναι απαραίτητο να αφαιρέσουμε από τα κράτη-μέλη αρμοδιότητες ε, και να έχουμε ενιαίο οργανισμό για την έγκριση τύπου όλων των οχημάτων. Δεν ε, χρειαζόμαστε, πιστεύουμε, επανάσταση. Αυτοί που σήμερα εγκρίνουν ε, τους τύπους ε, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι υπάρχει ανεξάρτητος φορέας ελέγχου που τους ελέγχει και σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων θα πρέπει να εφαρμόζονται κυρώσεις. Το Συμβούλιο, όπως γνωρίζετε, Εξαρτάται από την πολιτική βούληση για αλλαγή. Αυτό είναι πολιτικό θέμα. Ε, εγώ όμως θα ήθελα να ασχοληθώ ε, περισσότερο με το τεχνικό επίπεδο. Ο οργανισμός θα πρέπει να έχει επαρκείς αρμοδιότητες και θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να επιβάλλει κυρώσεις. Εάν απλά αξιολογεί χωρίς να μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις, αυτό δεν θα έχει νόημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να δώσω το λόγο στην Κριστίν. Κύριε Υπουργέ, Είπατε πολλάκις ότι τα οικονομικά ζητήματα, τα ζητήματα κόστους είχαν οδηγήσει σε κάποιες επιλογές. Είπατε ότι για να μειωθεί το δεξίδιο του άνθρακα ε, από οικονομικής πλευράς ήταν πιο συμφέρον αυτό αλλά τελικά είχαμε αύξηση του διοξιδίου του άζωτος. Εάν δείτε όμως την έκθεσή μας, ιδιαίτερα εκεί που αναφέρουμε τα συγκεκριμένα γεγονότα και τα συγκεκριμένα στοιχεία, δεν υπάρχει καμιά ε, αντινομία, καμιά αντίθεση ανάμεσα στη μείωση του διοξυδίου του άνθρακα και του αζότου. Ε, επίσης είπατε ότι το ντίζελ γενικά το προτιμούν οι καταναλωτές επειδή είναι πιο φτηνό. Φαντάζομαι ότι έκτοτε θα έχετε αυξήσει το, τη φορολόγηση του ντίζελ έτσι ώστε οι καταναλωτές να μην θεωρούν ότι είναι οικονομικό το να, ακολουθεί να, να προτιμά τον δίζελ όταν τελικά δεν είναι καθόλου οικονομικό ούτε καν για αυτούς για την υγεία του στο μέλλον. Τι έχετε κάνει λοιπόν σε ό,τι αφορά τα κίνητρα ή τα αντικίνητρα για τη χρησιμοποίηση του δίζελ ως καύσιμο. Ποια είναι η κατάσταση σε ό,τι αφορά τη ρήπανση ε, στη Σλοβακία. Εγώ είμαι Γαλλίδα ε, ζήσαμε και εξακολουθούμε να ζούμε ένα χειμώνα εξαιρετικά ρηπογόνο και για τα σωματίδια και για το δεξιό του άνθρακα και για το άζωτο. Ε, μιλάμε για το σήμερα, δεν μιλάμε για το αύριο. Φαντάζομαι ότι έχετε και στις ανησυχίες. Ε, ποια είναι η δική σας εκτίμηση και ποιες πολιτικές εφαρμόζεται σε επίπεδο ρύθμισης οικονομικής για τα διάφορα, μορφές καυσίμων να, να σας κάνω όλα τα ερωτήματά μου τώρα και για την απασχόληση. Ε, διότι βεβαίως οι αυτοκινητοβιομηχανίες είναι πολύ ενεργές στην χώρα σας. Φαντάζομαι ότι συζητήσατε με τις εταιρείες αυτές, έτσι ώστε οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται στα εργοστάσια τους να μπορέσουν να ε, εργαστούν, ε, να καταρτιστούν και να μπορέσουν να εργαστούν κάπου αλλού στο μέλλον πολλοί αλλάζουν, πολλοί αυτοβιομηχανίες αλλάζουν ε, τον τρόπο παραγωγής. Θα πρέπει λοιπόν ε, οι εξειδικευμένοι εργάτες, ε, εργαζόμενοι σας να επανακαταρτιστούν. Θα ήθελα και από αυτού κάποια στοιχεία. Ευχαριστώ. Θα αναφερθώ πρώτα στο περιβάλλον, πρωτού αναφερθώ στα όσα έχουμε κάνει ως χώρα. Ευτυχώς ε, δεν βρισκόμαστε στη θέση της Γαλλίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό το θέμα αυτό. Είμαστε μικρή χώρα και πιο ευέλικτη. Πάντα προσπαθούσαμε να ενεργούμε προορατικά όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. Γι' αυτό προτιμούμε τα αυτοκίνητα με, με μικρότερο κυβισμό. Κάτι ανάλογο ισχύει και για τα φορτηγά. όσον αφορά τη χρήση των αυτοκινητοδρόμων, για παράδειγμα. Θέλουμε να δώσουμε κίνητρα στους καταναλωτές να σκέφτονται με σύγχρονο τρόπο κατά την αγορά αυτοκινήτων ε, και εάν επιλέξει κανείς αυτοκίνητο με μεγάλο κυβισμό να πληρώσει ανάλογα. Οι καταναλωτές μας πάντως ε, γενικά δείχνουν ανάλογα ενδιαφέροντα με αυτά ε, καταναλωτών ε, σε άλλες χώρες. Όπως σας είπα, η έγκριση τύπου των οχημάτων ε, δεν γίνεται στη δική μας χώρα. Ε, στην χώρα μας ε, τώρα θα εγκατασταθεί και η Jaguar Land Rover. Ε, αυτό βέβαια είναι θέμα που αφορά κυρίως τις εξαγωγές. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα κλάστερ κατασκευαστών και να δημιουργήσουμε και ανάλογα κέντρα ερευνών στη Σλοβακία για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για λιγότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος και αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Η Σλοβακία ε, θέλει να βασίζεται και στο εργοτικά δυναμικό. Έχουμε εισάγει διτό σύστημα ε, ε, κατάρτισης και εξηγούμε στους πολίτες μας ε, τι σπουδές συμφέρει να κάνει κανείς, ε, σε ποιους τομείς μπορεί να ε, έχει καλή ευκαιρία για θέση εργασίας. Θέλουμε έτσι να δημιουργήσουμε προστιθέμενη αξία εντός της Σλοβακίας. Αυτό με την ανάπτυξη της ρομποτικής θα είναι θετικό για το μέλλον. Και θα μας βοηθήσει να επενδύσουμε στην ανάπτυξη και να κοιτάμε το μέλλον. Eh, Ο κύριος Γερμπράντη έχει το λόγο. Όχι, δεν θέλετε το λόγο. Πολύ ωραία. Πάμε στον επόμενο μιλητή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, Να δούμε τι θα γίνει τώρα με το Brexit με και τις αγγλικές εταιρείες, τις βρετανικές. Από τη δική σας προοπτική μπορεί να είναι πιο εύκολο Εσείς στο Συμβούλιο πώς το βλέπετε πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη ευρωπαϊκή επιρροή σε εθνικό επίπεδο V prvom rade na, na odľahčenie. Samozrejme, my sme vďační za príchod e, Jaguaru Land Καταρχάς, να πω ότι χαιρόμαστε πολύ που ε, έρχεται σε μας η Land Rover. Είναι ε, η τελευταία επένδυση στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία 7 χρόνια. Και μέχρι τελευταία στιγμή ανταγωνιζόμασταν με το Μεξικό για, ε, για αυτή την εγκατάσταση. Αυτό είναι πολύ θετικό, όχι μόνο για τη Σλοβακία. Όσον αφορά το δεύτερο τμήμα της ερώτησής σας. Στο Συμβούλιο δύο φορές συζητήθηκε, μία φορά τον Ιούνιο και μία φορά τον Δεκέμβριο. Κατά την ε, Ολλανδική Προεδρία δηλαδή και κατά την Σλοβακική Προεδρία. Υπήρξε συμφωνία σε επίπεδο Συμβουλίου ότι πρέπει να εφαρμόσουμε καλύτερα τους ισχύοντες κανόνες και ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε τους ισχύοντες κανόνες. Αυτές είναι οι βασικότερες πτυχές. Επίσης συζητήθηκε η απαγόρευση των συστημάτων αναστολής. Και υπήρχε συμφωνία στο Συμβούλιο ότι χρειαζόμαστε νέα εποπτεία αγοράς υπό τη μορφή ε, νέου οργανισμού. Αυτές είναι οι συζητήσεις που έγιναν σε επίπεδο Συμβουλίου. Θα συνεχιστούν οι συζητήσεις. Και χάρη σε εσά, χάρη στο Κοινοβούλιο δηλαδή. Και χάρη στις εργασίες της Επιτροπής σας. Έχετε εκπονήσει πολύ καλά έγγραφα, τα οποία θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο γνωρίζει τώρα ποια είναι η θέση σας. και πού μπορεί να βασίζεται στην υποστήριξη του Κοινοβουλίου. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι θεωρούμε την Επιτροπή σας πολύ καλό φορέα για την επικοινωνία στο θέμα αυτό. Αποτελεί πολύ καλή αρχή. Είναι θετικό το ότι οι ευρωβουλευτές συμμετέχουν ε, ήδη από την αρχή στη νέα διαδικασία. Τα κράτη-μέλη έτσι έχουν τη δυνατότητα να μάθουν ε, τις θέσεις ε, των άλλων ευρωβουλευτών και κρατών μελών. Ευχαριστώ. Έχω άλλο ένα ερώτημα. Πώς εξηγείτε αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι δηλαδή οι καταναλωτές, ε, οι άνθρωποι και στην Σλοβακία και στις κάτω χώρες ε, δεν φαίνεται να έχουν επηρεαστεί τόσο πολύ ε, για το σκάνδαλο αυτό. Ξεκολουθεί δηλαδή να, πουν, να αγοράζουν ε, κάποια μοντέλα. Βλέπω ότι είστε μηχανικός ε, στο βιογραφικό σας. Πρέπει να θέτουμε όμως και πολιτικά ζητήματα. Τι συμβαίνει τελικά. Zareagovať na to je asi najlepším Πρέπει να σας δώσω νομίζω ε, ένα παράδειγμα. Ας πάρουμε μια άλλη εταιρεία στον τομέα της επικοινωνίας. Η Samsung δημιούργησε ένα νέο προϊόν, περίμενε τεράστια κέρδη αλλά τελικά αυτό το νέο προϊόν δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ούτε καν σε, στα αεροπλάνα. Θα έπρεπε λοιπόν και πάλι να επανεξετάσει το θέμα, να πείσει τους καταναλωτές. Στην πολιτική, λοιπόν, βλέπει κανείς εάν έχει πείσει τους ψηφοφόρους ή όχι. Μια επιχείρηση που έχει χάσει την εμπιστοσύνη των, πολι... των καταναλωτών έχει να αντιμετωπίσει δύο θέματα. Καταρχάς την πτώση των μετοχών. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί πια να λειτουργήσει η επιχείρηση. Αυτό φαίνεται άλλωστε από τις τιμές των μετοχών. Το δεύτερο πρόβλημα είναι η εμπιστοσύνη των πελατών. Οι καταναλωτές νιώθουν ότι έχουν εξαπατηθεί και αυτό φαίνεται ε, στις πολίτες των διαφόρων προϊόντων. Αυτά τα σημάδια μειωμένης ενοχής αποτελούν θετικά στοιχεία και όσον αφορά την Samsung που ωστόσο ξεπέρασε την κρίση με πολύ θετικό τρόπο. Νομίζω ότι έμαθε ο τομέας από το σκάνδαλο αυτό και Τελικά όλα αυτά ωφελούν τους καταναλωτές, τους οδηγούς αυτοκινήτων, που είναι πιο ενημερωμένοι κατά την αγορά οχήματος. Αυτό επίσης ωφελεί και το περιβάλλον. Ευχαριστώ και ο Σέπτανς για ένα εξάλεπτο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ με τον κύριο Βαντερκάμπ. Uh, για το Brexit. Θα γίνει πολύ πιο ελκυστικός προορισμός για τις βρετανικές επιχειρήσεις στη Σλοβακία από τη Βρετανία. Μια τραγωδία που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Δώσατε κάποιες ενδείξεις. Είπατε ότι θα υποστηρίξετε την ιδέα ευρωπαϊκής εποπτείας. Υπάρχει κάποιο θέμα όμως ερωτηματικό για το επίπεδο των ευθυνών. Εκφράστε ανησυχίε γι' αυτό. Κάποια σχόλια κάνατε, να μην επαναληφθούν αυτά που γίνονται, που γίνονται σε άλλα μέρη του κόσμου, είπατε, γιατί ίσω να μην ενδείκνεται ω μέτρα εδώ, το κατανοώ αυτό. Αλλά η διαδικασία εκμάθηση από τι βέλτιστε πρακτικέ είναι αμφίδρομη διαδικασία. Εμεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση περιμένουμε από άλλου να προσαρμοστούν και να μάθουν από πολιτικέ που είναι σωστέ εδώ. Και εκεί που κάνουμε λάθη, σίγουρα θα θέλαμε να προσαρμοστούμε και να μάθουμε από άλλου. Ποια στοιχεία γραφειοκρατικού άχθου είναι αυτά που αναφέρεται στην απάντηση στην ερώτηση 1. Ποια στοιχεία γραφειοκρατικού άχθους σα προβληματίζουν για τις ενδεχόμενε ευθύνε εποπτική αρχή ευρωπαϊκής. Ποιε είναι οι βασικέ σα ανησυχίε. Τι μα ζητάτε να αποφύγουμε. E, Όσον αφορά το διοικητικό άχθος και τη γραφειοκρατία, μία πρόταση θα σας πω. Κανένας οργανισμός δεν έχει νόημα εάν δεν έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Νόημα έχει όταν έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες, όταν φέρει ευθύνη και όταν ε, μπορεί να εφαρμόσει κάποια πράγματα. Αλλιώς δεν έχει κανένα νόημα. Εάν ένας οργανισμός διαπιστώνει προβλήματα στην πράξη όμως δεν έχει τη δυνατότητα να διορθώσει ε, τα προβλήματα, τότε δεν έχει κανένα νόημα η ύπαρξη ενός τέτοιου οργανισμού. η αύξηση του διοικητικού άχθους δεν αποτελεί και τραγωδία κατά τη δημιουργία νέου οργανισμού εφόσον βοηθήσει στην πράξη αυτό, εφόσον υπάρχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Η Σλοβακία συμφωνεί με τη δημιουργία ενός τέτοιου οργανισμού μόνον εφόσον είναι οργανισμός με συγκεκριμένες αρμοδιότητες και με τη δυνατότητα να κάνει κάποια πράγματα στην πράξη. Αναφέρθηκαν ε, και οι ε, ε, αξιολογήσεις ομοτήμων, peer reviews, αμοιβαία αξιολόγηση μεταξύ των κρατών μελών ή ανταλλαγή ε, των αξιολογήσεων. Θα μπορούσε αυτό να αποτελέσει μέρος μιας λύσης, μόνο όμως μέρος μιας λύσης. Πρέπει να εφαρμόζουμε ενιαία πρότυπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να αξιολογείται και η παροχή υπηρεσιών. Είναι σημαντικό να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για όλους κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας. Προτείναμε μία διαδικασία ε, επιστοποίησης ε, για τους παρόχους υπηρεσιών. Ευχαριστώ. Φαίνεται να διαφαίνεται μια συνένεση ότι χρειάζεται αποτελεσματική εποπτεία και προφανώς πρέπει να διεξαχθεί πολιτική συζήτηση από αυτού. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία που εντάσσονται στη διαδικασία. Η έγκριση τύπου και η σχετική διαδικασία εξετάζεται σε μια άλλη επιτροπή. Έγιναν διάφορες προτάσεις από την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Διερωτώ με, ποια είναι η άποψή σας επ' αυτόν. Κατανοώ ότι μπορεί να μην έχετε άποψη για τα πάντα, αλλά ίσως να έχετε κάποιες ιδέες γενικές. Πρώτα απ' όλα, εθνικό σύστημα τέλους για τη χρηματοδότηση έγκριση τύπου που θα πληρώνεται από τον κατασκευαστή που κάνει αίτηση για έγκριση τύπου και θα καθορίσετε το τέλο από κάθε κράτο μέλο ξεχωριστά. Να μην υπάρχει εμπορικό δεσμό μεταξύ κατασκευαστού τεχνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εγκρίσεω τύπου. Έχετε άποψη από αυτό. Δεύτερον, εθνικό τέλο 10 ευρώ ανά όχημα που πωλείται για να χρηματοδοτείται η εποπτεία και θα πρέπει επίσης να υπάρχει και ανταλλαγή πληροφοριών για υποπτή σε κάθε και ανεξάρτητη επιτροπή ελεγκτών που ελέγχουν τις αρχές εγκρίσεως τύπου των κρατών μελών. Εντάξει, μακροσκελής κατάλογος στο διαθέσιμο χρόνο. Έχετε κάποια άποψη από αυτόν. Θα σας είμαι θα ευγνώμονες αν έχετε άποψη από αυτόν. Ε, ten, ε, ten zoznam bol pomerne dlhý, s kolegami sme ναι, είναι μακροσκελής ο κατάλογο και το έχουμε συζητήσει επανειλημμένα με του συναδέλφου μα. Όλα τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο συμφώνησαν να μην πληρώνει ο κατασκευαστής τον ε, ελεγκτή, αλλά αυτό είναι δύσκολο να εφαρμοστεί στην πράξη και όσον αφορά το μέλλον. Για μας έχει περισσότερο νόημα να ακολουθήσουμε το δρόμο της ενίσχυσης ε, των ελέγχων. Και ακριβώς αυτό θα πρέπει να υποπτεύει ο οργανισμός. όσον αφορά την ελεγκτική ομάδα. Συμφωνώ μαζί σας. Και ήδη το τόνισα επανειλημμένα σήμερα όσον αφορά τη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και ως έκχροντ μπορεί να κλείσει αυτό το γύρο. Ναι, σας ευχαριστώ για την αφορά. Να δούμε λίγο και το μέλλον. Μια από τις ε, σημαντικές συζητήσεις που θα γίνουν θα αφορούν το τέταρτο πακέτο RDE έχει να κάνει με την, την συμμόρφωση ε, in service. Στις ΗΠΑ τη στιγμή κάνουν τεστ έκπληξη, ευνηδιαστικούς ελέγχους. Εμείς επειδή δεν εμπιστευόμαστε οι μένοι τους δε χώρες, ε, θέλει ο καθένας να δει τι τεστ θα του προτείνει ο άλλος, έτσι λοιπόν όποιο τεστ ε, αποφασίσουμε είναι γνωστό στην κάθε λεπτομέρεια. Δηλαδή ξέρει ο κατασκευαστής πώς θα λεφθεί το αυτοκίνητό του. Οι Αμερικανοί λοιπόν λένε ότι αυτά τα οποία, αυτό που είναι κρίσιμο είναι ένα τεστ έκπληξη. Ένα τεστ για το οποίο να μην έχουν προετοιμαστεί οι αυτοκινητοβιομηχανίες. Ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό. Jasné. Καταρχάς, θα ήθελα να πω ότι η Σλοβακία εμπιστεύεται τις χώρες που εγκρίνουν τα αυτοκίνητα. Δεν λέμε ότι εμείς φτιάχνουμε καλά αυτοκίνητα ή άλλοι εφαρμόζουν κακές δοκιμές. Όχι, λέμε ότι πρέπει να αλλάξει το σύστημα και να δημιουργήσουμε κανόνες για να αποφύγουμε παρόμοιες καταστάσεις. Όσον αφορά τις ευνηδιαστικέ δοκιμές, ε, αυτές εφαρμόζονται και στον αθλητισμό, όπου έχουν βελτιωθεί πολύ τα πράγματα. Βλέπουμε λιγότερα περιστατικά ε, ντόπινγκ και κάτι παρόμοιο θα οδηγούσε και τον τομέα των αυτοκινήτων. Αυτό βέβαια θα εξαρτηθεί από την ε, μόρφη που θα λάβει η νομοθεσία γενικά και από την εφαρμογή της. Κατά τη σύγκριση της ε, κατανάλωσης αυτοκινήτων μάλιστα του ιδίου αυτοκινήτου υπό παρόμοιες ε, συνθήκες, βλέπουμε πάλι να υπάρχουν διακυμάνσεις ε, διότι ε, επηρεάζει την κατάσταση, ο καιρός, οι συνήθειες του οδηγού κλπ. αλλά θα είναι χρήσιμο να έχουμε ελέγχους που να βασίζονται σε παρόμοιους παράγοντες. Θα πρέπει όμως να καταλήγουμε σε δοκιμές με μόνο σήμαντα αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Ένα τελευταίο σχόλιο την πλευρά μου. Όλες οι αρχές έγκρισης τύπου σίγουρα έκαναν τα τεστ όπως προβλεπόταν, αλλά ήξεραν ακριβώς οι αυτοκινητομηχανίες πώς θα ελεγχθούν τα αυτοκίνητα και μπορούσαν να κάνουν διάφορα κόλπα. Μετά από τα 22 λεπτά, ας πούμε, μπορούν να μειώσουν τις, ε, ε, να, να αποσύρουν τα μηχανήματα εκπομπών. Ενώ το τεστ κρατάει 20 λεπτά. Γι' αυτό λοιπόν είναι, έχει σημασία είναι σημασία να μπει στη συζήτηση το θέμα του τεστ έκπληξη σε ό,τι αφορά το in-service conformity. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. μιλάμε για μη αποτελεσματική εποπτεία την οποία θα πρέπει να αλλάξουμε. Και ακριβώς γι' αυτό καταβάλλονται κοινέ προσπάθειες για τα ελαφρά οχήματα να εφαρμόσουμε ενιαία διαδικασία. κάτι που θα ωφελήσει και τους καταναλωτές και το περιβάλλον. Ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η ακρόαση να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τις συνεισφορές τους αλλά και τον Υπουργό για την εξαιρετικά χρήσιμη και ενδιαφέρουσα αυτή ακρόαση. Όποιος θέλει να υποβάλει περαιτέρω ερωτήματα γραπτός μπορεί να απευθυνθεί στη γραμματεία έως τις 19 Ιανουαρίου. Θα διακόψουμε τώρα έως τις 3.